Καλημέρα αγαπητοί συνάδελφοι. Τέσσερις φορές έχουμε πει σήμερα. Καλημέρα. Την πέμπτη θα με κεράσετε καφέ. Αστείευεται η πρόεδρος. Μπορούμε να ξεκινήσουμε. Θα ήθελα να συζητήσω πρώτα απ' όλα στη μνήμη του Προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας, του Ζακ Σιράκ, ο οποίος πέθανε στις 25 Σεπτεμβρίου του 2019 και ήταν και μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και μέλος της, Ευρωπα... Ε, Επιτροπής Μεταφορών το 79 μέχρι τον Απρίλιο του 80. Θα ήθελα λοιπόν στη μνήμη του Ζακ Σιράκ να σας ε, ζητήσω να τηρήσουμε ενός λεπτού σιγή. Je vous remercie, mes chers collègues. Ευχαριστώ. Sans plus perdre de temps. Λοιπόν, χωρίς να καθυστερούμε. εδώ μπορούμε να εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη. Σας ευχαριστώ. Μπορούμε να εγκρίνουμε τα πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης, των προηγούμενων συνεδριάσεων, αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις. Σας ευχαριστώ. Τώρα, θα ήθελα να σας προσκαλέσω να σας ενημερώσω για το ημερολόγιο σας στις 3 Δεκεμβρίου. Σας προσκαλώ όλα τα μέλη της ε, Επιτροπής μας, καθώς επίσης και τους συνεργάτες σας και τους βοηθούς σας. Είναι και τελευταίος μήνας, ο Δεκέμβριο τον οποίο θα μπορέσουμε να κάνουμε αυτή την ε, μικρή εκδήλωση. Να σας προσκαλέσω λοιπόν στις 3 Δεκεμβρίου στη διεξίωση εν ώψη των γιορτών των Χριστουγέννων στις 6 ώρα το απόγευμα, δηλαδή μετά την συνεδρία της Επιτροπής μας. Λογικά θα Έχουμε το νέο Επίτροπο Αρμόδιο για θέματα μεταφορών και καθώς επίσης και εκπροσώπηση από τη Φινλανδική Προεδρία στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα λάβετε και ε, γραπτός ε, την πρόσκληση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ας περάσουμε τώρα στις εκλογές. Αγαπητοί συνάδελφοι, όπως γνωρίζετε θα πρέπει να εκλέξουμε τους ε, δύο αντιπροέδρους μας, τον πρώτο και τρίτο αντιπρόεδρο της Επιτροπής μας, μετά από τις παρετήσεις των κυρίων Ντάνιελσον οποίος ε, ε, παραιτήθηκε προκειμένου να γίνει συντονιστής της ομάδας των συντονιστών και του κυρίου α, Ουλεγή. Θα πρέπει λοιπόν να εκλέξουμε τον πρώτο και τον τρίτο αντιπρόεδρο. Για την θέση του πρώτου αντιπρόεδρου οι ε, σοσιαλιστές και δημοκράτες μας έχουν προτείνει τον κύριο Ολύρη και θα ήθελα να ρωτήσω εάν υπάρχουν άλλες υποψηφιότητες εκτός από εκείνη του κυρίου Ούγελη. Από ό,τι φαίνεται. Όχι, οι σοσιαλιστές και οι δημοκράτες συνεχίζουν να υποστηρίζουν την κυριό Ούγελη. Κύριε κύριος Τάνελσον απαντάει ναι. Κύριε Ούγελη, εσείς. Ένα λεπτό. Πρώτα απ' όλα συμφωνείτε, πρέπει να σας ρωτήσω. Εάν δεν υποβάλλεται άλλη υποψηφιότητα, δεν χρειάζεται να κάνουμε μυστική ψηφοφορία. Μπορούμε να προχωρήσουμε σε εκλογή διαβοής. Συγχαρητήρια κύριε Ούγελη. Ε, έχετε εκλεγεί πρώτος αντιπρόεδρος. Μπορείτε να έρθετε στο Προεδρείο. Μπορούμε να συνεχίσουμε. Ελάτε, ελάτε. στην εκλογή. Του τρίτου αντιπροεδρού της Επιτροπής μας. Να μην ζηλεύετε. το τρίτο λοιπόν Αντιπρόεδρου. Οι σοσιαλιστές και οι δημοκράτες μας έχουν προτείνει τον κύριο Άμεριξ ως υποψήφιο για τη θέση του τρίτου αντιπροέδρου. Οι σοσιαλιστές ε, συνεχίζουν να υποστηρίζουν την υποψηφιότητα. Ο κύριο Ντάνιλσον απαντά ναι. Θα ήθελα να ρωτήσω αν κάποια άλλη πολιτική ομάδα θέλει να αποβάλει άλλη υποψηφιότητα. Ο κύριος Ολιβιέ από την ομάδα ID προτείνω την κυρία Λεσοντέ και ζητώ να γίνει μυστική ψηφοφορία. Κυρία Λεσοντέ, συμφωνείτε με το να είστε υποψήφια. Εκτός μικροφώνου. Κύριε Άμεριξ, πού βρίσκεστε. Δεν σας είχα το συγγνώμη. Ε, συμφωνείτε και εσείς με την υποβολή της υποψηφιότητά σας, σα ρωτώ. Ναι, απαντάει ο κύριο Σάμαριξ. Ωραία. Θα προχωρήσουμε λοιπόν σε ηλεκτρονική ψηφοφορία, μια και ζητήθηκε. Θα ήθελα να ε, εξασφαλίσουμε πρώτα όλα όσα προβλέπει ο κανονισμός. Ε, πρώτα απ' όλα να ελέγξουμε την απαρτία. Βάλτε την κάρτα σας στο, στο μηχάνημα, ψηφίστε παρακαλώ για να ελέγξουμε την απαρτία. Είναι τέστα τώρα, δεν ψηφίζουμε για τον Αντιπρόεδρο. Μπορείτε να ψηφίσετε ό,τι θέλετε, απλώς θέλω να ελέγξουμε αν έχουμε την απαρτία. Ωραία. Έχουμε απαρτία. Alors, comme euh, μια και είναι αυστηρή διαδικασία που ακολουθούμε, θα πρέπει να διαβάσω τα ονόματα των ε, τακτικών μελών που στην ψηφοφορία θα αντικαταστήσει κάποιο ο αναπληρωματικό. Ο κύριο Σούλτ από το ΕΛΚ ε, αντικαθίσταται από τον κύριο Γκάλερ. Είστε εδώ. Καλημέρα. Κυρία Κουζένσκα, αντικαθίσταται. Αντικαθίσταται τον κύριο Φροκόφσκι. Είστε εδώ. Ευχαριστώ. Κυρία Μοντέρο, από τον κύριο Ναμπούκοφ. Ναβόκοφ, συγγνώμη. Κύριος, είστε, ε, κύριε Ναβόκοφ, είστε εδώ. Καλημέρα, ευχαριστώ. Euh, Ξέρετε, καμιά φορά πρέπει να τα ελέγξουμε όλα, κύριε Μαρινέσκου. Για τους σοσιαλιστές, η κυρία Κραπίνη, είστε εδώ. Για τους πράσινους, κύριο Έσλι. Από, την κυρία Ντόνιγκ αντικαθίσταται. Είστε παρούσα. Καλημέρα. Κυρία Τίλιμετς. Αντικαθίσταται και την κυρία Εύανς. Καλημέρα. Και η κυρία Βόζενμπερκ. Από την κυρία Μπίρκινεν. Είστε παρούσα. Και ο κύριος Μελασσό. τον κύριο Φέρπερ. Και ακόμα. Κυρία Λέιλα μπει καλημέρα. Έχετε το λόγο. Αντικαθιστώ την κυρία Κονέσινα. Η πρόεδρος χωρίς μικρόφωνο δυστυχώς μιλάει. Δεν την ακούμε. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Σας ε, είχα ξεχάσει. Και ο κ. Φλέγκο με την κυρία Νάν Κιβάλ. Ο κύριος Φλεγκό είναι εδώ. Ψηφίζετε κύριε Φλεγκό. Κύριε Μαρινέσκου, θέλετε το λόγο. Η κυρία Βίρκονεν αντικαθιστά την κυρία Βόζεμπερ. Το είπατε. Α, συγγνώμη, συγγνώμη. συγγνώμη. Κύριε Μαρινέσκου, δεν θέλετε να έρθετε εδώ πάνω και να κάνετε τη δουλειά μου. Όχι, έμε ε, τίποτα. Το φανταζόμουν. Ωραία. Συνεχίζουμε με τη διαδικασία. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Μυστική ψηφοφορία λοιπόν. Έχουμε δύο υποψήφιους. Το πράσινο είναι για τον κύριο Άμεριξ. Το πράσινο, επαναλαμβάνω, για τον κύριο Άμεριξ. Και το κόκκινο για την κυρία Λεσόντε. Και αν δεν έχετε προτίμηση πατάτε το άσπρο, που είναι η αποχή. Οι εποχές δεν μετράνε. Εντάξει, το πράσινο κουμπί για τον κύριο Αμερίξ, το κόκκινο για την κυρία Λεσόντε. Είστε έτοιμοι? Κύριε Ρικέ, είστε έτοιμος? Κύριε Ρικέ, μα επιτρέπετε να συνεχίσουμε. Ωραία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πράσινο για τον κύριο Άμεριξ, κόκκινο για την κυρία Λεσοντέ. Le vote est Λίγη ψηφοφορία. Ο κύριος Άμεριξ εκλέγεται με 34 ψήφους κυρία Λεσόντε πήρε εννέα ψήφους. Κυρία Μερίξ, παρακαλώ πολύ μπορείτε να έρθετε εδώ μαζί μας ως τρίτος αντιπρόεδρος της Επιτροπής μας. Συγχαρητήρια. Allez, sans Περνάμε στα σημεία 6 και 7. Πρόταση απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που δίνουν την άδεια στη Γερμανία να τροποποιήσει την υπάρχουσα διμερή συμφωνία για χερσές μεταφορέ με την Ελβετία προκειμένου να επιτραπεί το καμποτάζ ε, στις για τις μεταφορές με πούλμαν και λεωφορεία στις ε, μεθόρειες, παραμεθόριες περιοχές των δύο χωρών. Εισηγητής ο κ. Φέρμπερ. Είναι δύο οι προτάσεις που έχουμε συγκεκριμένα. Η μία είναι για τη Γερμανία, η άλλη είναι για την Ιταλία. Προκειμένου να τροποποιήσουν τις ε, διμερείς συμφωνίες με την Ελβετία. Και οι δύο αυτές εκθέσεις έχουν τον ίδιο εισηγητή, και τους ίδιους και ηγητές. Θα τη συζητήσουμε τώρα αμέσω. Δίνω το λόγο στον κύριο Φέρμπερ για πέντε λεπτά. Μετά θα δώσω το λόγο στους κοιόδης ηγητές και θα ζητήσω από τον κύριο Φέρμπερ να κλείσει. Πέντε λεπτά ο λόγος του κύριο Φέρμπερ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, θα είμαι και πιο σύντομος ελπίζω. Είναι σημαντικό βεβαίως το θέμα αφορά και την χώρα μου, δεν είναι όμως τόσο περίπλοκο. Μέσω αυτών των εκθέσεων εξουδοτείται η Ιταλία να συνάψει συμφωνία καμποτάς με την Ελβετία και από την άλλη η Γερμανία η οποία έχει ήδη υφιστάμενη τέτοια συμφωνία για τις διασυνοριακές ε, συγκοινωνίες να την επεκτήσει. Αυτά περιορίζονται στις μεθοριακές περιοχές. Στόχος είναι να βελτιωθεί οι, διασυνο... να διασυνο... οι δημόσιες διασυνοριακές μεταφορές, κατά το οποίο θα ωφελήσει τους εργαζόμενους στις μεθοριακές περιοχές και στις δύο κατευθύνσεις. Ο λόγος είναι πως από όταν ε, ε, τέθη ενισχύ η συνθήτης της ε, Λισαβόνας αυτά είναι κοινοτική αρμοδιότητα. Υπήρχαν όμως για ιστορικούς λόγους μια συμφωνία μεταξύ της Γαλλίας και της Ελβετικής ε, Συνομοσπονδίας ε, και της Γερμανίας. Τώρα θα προσαρμόσουμε τη Γερμανική Συμφωνία και οι Ιταλοί θέλουν επίσης να διαπραγματευτεί μια τέτοια συμφωνία και άρα πρέπει να τους δώσει την δυνατότητα η Ευρωπαϊκή Ένωση να το κάνουν διμερός. Οπότε Αυτά αφορούν ε, την ίση μεταχείριση των σχετικών επιχειρήσεων και δεν θα υπάρξει έβριση του ανταγωνισμού. Πρόκειται για την δυνατότητα που πρέπει να δοθεί στις χώρες, οπότε δεν έχουμε να συζητήσουμε κάπου, κάτι επί της ουσίας. Απλά εξοδότηση για να γίνουν αυτές οι διαπραγματεύσεις. Το Συμβούλιο ε, δυστυχώς είναι κάπως πιο γρήγορο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά δεν είχε και εκλογές βεβαίως όπως εμείς, οπότε ήδη αρχές Ιουλίου αποφάσισε και υπάρχουν μόνο γλωσσικές και νομικές αλλαγές ε, στο κείμενο και εγώ δεν βλέπω κάποια ανάγκη για ουσιαστικές ε, τροπολογίες. Ε, έχω υποβάλει μόνο μία για την νομική βάση, την οποία δέχτηκε και το Συμβούλιο, κάτι το οποίο βέβαια σημαίνει ότι πρέπει να εμπλακεί και η Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων του Κοινοβουλίου. Ε, κατά κανόνα βεβαίως αυτό γίνεται γρήγορα υπό μορφή επιστολής. Ελπίζω λοιπόν να συμφωνήσουν με τον εισηγητή και το Συμβούλιο, αν και εγώ δεν είμαι νομικός και γνωρίζω ότι αυτά τα πράγματα με τους νομικούς είναι πάντα επικίνδυνα. Γι' αυτό η πρότασή μου είναι απλά να υπάρξει μια αλλαγή της νομικής βάσης και θα ήθελα να πάμε σε μια απλοποιημένη διαδικασία γρήγορα με το Συμβούλιο έτσι ώστε οι δύο χώρες που θέλουν να ξεκινήσουν αυτές τις διαπραγματεύσεις να το κάνουν. Λοιπόν, τρία λεπτά τελείωσα. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Ντάνιελσον για τους ε, σοσιαλιστές. Ε, ευχαριστώ. Θα μιλήσω σου ειδικά. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για το έργο του. Όπως είπε και εκείνος, το θέμα είναι πολύ σημαντικό, αλλά δεν είναι περίπλοκο. Είναι σημαντικό για τις θέσεις εργασίας, είναι σημαντικό για την εσωτερική αγορά και για την οικονομική ανάπτυξη. Είναι σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη της να έχουν καλές σχέσεις με τις όμορες χώρες. Ιδιαίτερα με αυτές, με μια χώρα όπως η Ελβετία που βρίσκεται ε, που έχει κοινά σύνορα με τη Γαλλία, με τη Γερμανία, με την Ιταλία. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε ε, αποτελεσματικές μεταφορές ε, με λεωφορεία. Αυτό εξυπηρετεί την καθημερινότητα των πολιτών που ζουν στις μεθοριακές περιοχές. Σύμφωνα λοιπόν με τον εισηγητή θα πρέπει αυτές οι συμφωνίες να συναυθούν όσο το δυνατόν πιο σύντομα και να φροντίσουμε να μην υπάρξει διακριτική μεταχείριση εις βάρος κάποιων ε, επιχειρήσεων κάποιων ε, και να μην δημιουργηθούν σταρβλώσεις στον ανταγωνισμό. Για το ε, Renew, κύριος Πάος Δαντίας. Θα συνεχίσω στα ισπανικά. Το πρώτο που θα ήθελα να πω, πρώτα απ' όλα να συγχαρώ τον εισηγητή. Πιστεύω ότι και οι δύο αυτές προτάσεις για να επιτραπεί η σύναψη συμφωνίων καμποτάζ είναι πολύ ενδιαφέρουσες και επίσης να τονίσω ότι είναι πολύ σημαντικό και οι δύο αυτέ συμφωνίε και για την Ιταλία και για την ε, Γερμανία να συνάδουν με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Είναι εύλογο. Επίσης, αυτές οι δύο συμφωνίες μεταξύ Γερμανίας και Ελβετίας και Ιταλίας ε, Ελβετίας να ε, εξασφαλίζουν την σωστή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, θα δώσουν δυνατότητες στους καταναλωτές αλλά και Στι ε, εταιρείε που δραστηριοποιούνται στο χώρο, να φροντίσουμε να μην, υπάρχουν, να μην υπάρχει διακριτική μεταχείριση ει βάρο των εταιριών τη ευρωπαικη ενωση Ευελπιστώ λοιπόν να ολοκληρωθεί αυτό το έργο πολύ σύντομα. Επόμενη σκιώδη συγγετρία είμαι η ίδια. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για το έργο σας. Το σημαντικό στο κείμενο αυτό είναι να δείξουμε και το φρόντισε αυτό ο εισηγητής, να δείξουμε ότι ο βασικός μας στόχος είναι να ενισχύσουμε τις διασυνοριακές μεταφορές μεταξύ Ελβετίας και Γερμανίας-Ταλίας, φροντίζοντας να μην υπάρξει κοινωνικό dumping. Γιατί ξέρετε ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό πρόβλημα. Ε, είναι ακριβώς αυτό που δημιουργεί προβλήματα στις, στις ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες. Ε, και αυτό που εγώ επισημαίνω, γιατί κατά τα άλλα συμφωνώ πλήρως με τον εισηγητή και υποστηρίζω την έκθεση του. 48 δευτερόλεπτα μου πήρε εμένα. Για το ID δεν έχουμε σκιώδη εισηγητή. Μήπως υπάρχει κάποιος που θα αντικαταστά, τον κύριο Καμπομενόζη. Εκτός μικροφώνου κάποιο σχόλιο. Εντάξει λέει η πρόεδρος. Για το ECR, Ρόμπερτ Σίλε. Όπως πάντοτε το ECR, όταν έχουμε έκθεση του κυρίου Φέμπερ, λαμβάνει υπόψη τις προτάσεις μας, συνέβη αυτό και εδώ. Ωστόσο, όσον αφορά την ουσία, νομίζω ότι δεν καλύπτεται παρκώς το κοινωνικό dump η Ελβετία θα επιδοθεί σε κοινωνικό ντάμπινγκ έναντι ε, κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επομένω, καλύπτεται παρκώς το θέμα και βεβαίως μπορούμε να υποστηρίξουμε την εκθέση του. Κύριε Κουντουρά, έχετε το λόγο για την ΚΟΕ. Θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή για τι δύο αυτέ προτάσει. Έχει κάνει πολύ καλή δουλειά και συμφωνούμε. Yeah. Θέλει κανείς άλλο το λόγο. Όχι. Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πού βρίσκεστε. Σας ε, βλέπουμε κάθε μέρα. Δεν μου είναι δυσάρεστο. Τι ευγενικό που είστε, λέει ο πρόεδρο. Έχετε το λόγο. Θα είμαι σύντομο. Να ευχαριστήσω τον εισηγητή που στηρίζει την πρόταση της Κομισιόν να δοθεί η άδεια στη Γερμανία και στην Ιταλία για αυτή τη διαπραγμάτευση. Να σας θυμίσω ότι υπάρχουν όροι οι οποίοι τίθενται προκειμένου η Γερμανία και η Ιταλία να προβούν σε αυτή τη διαπραγμάτευση. Η τελική συμφωνία δεν μπορεί να διαστρεβλώνει τον ανταγωνισμό και δεν μπορεί να γίνουν διακρίσεις ανάμεσα σε μεταφορής διαφορετικών χωρών. Ο εισηγητής είπε ότι γίνεται ακόμα συζήτηση για την νομική βάση. Η πρόταση Κομισιόν είναι το άρθρο 2 της Συνθήκης Ευρωπαϊκή Ένωσης και το άρθρο 91 για την τη συνθήκη για τη λειτουργία τη Ευρωπαϊκή Ένωση, διπλή νομική βάση. Είναι αλήθεια ότι υπάρχει το θέμα του άρθρου 2, του κατά πόσον αυτή η αναφορά στο άρθρο 2 είναι απαραίτητη. Περιμένουμε τη γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου. Το πιο σημαντικό είναι και δεν αμφισβητείτε ότι ε, η άλλη νομική βάση από την συνθήκη λειτουργία της Ευρωπαϊκή Ένωση θα παραμείνει. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Φέρμπερ, έχετε ξανά το λόγο για να κλείσουμε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα ευχαριστώ τους ε, συναδέλφους που ασχολήθηκαν με αυτό το όχι τόσο δύσκολο θέμα. Χαίρομαι για την συμφωνία που υπάρχει και να συμφωνήσω και με τον κύριο Τσίλε. Οπωσδήποτε δεν νομίζω να είναι θέμα το κοινωνικό dumping. Έχουμε κάποια άλλα προβλήματα στο θέμα του καμποτάζ, γιατί η Ελβετία είναι και στον χώρο Σέγγεν και υπάρχουν κάποια άλλα προβλήματα τα οποία θέλουν να λυθούν Γερμανοί και Ιταλοί γιατί είναι πολύ ε, διασυνδεδεμένη η αγορά εργασίας ε, και στις δύο πλευρές ε, των συνόρων. Θέλουμε λοιπόν να υπάρχουν ακριβώς οι δυνατότητες μεταφοράς με διασφάλιση των κοινωνικών δικαιωμάτων. Οπότε ε, πρέπει να προσέξουμε να μην παραβιαστεί το ευρωπαϊκό δίκαιο με αυτές ε, τις ε, διμερείς συμφωνίες και η Κομισιόν έχει όχι μόνο το δικαίωμα αλλά την υποχρέωση να παρακολουθήσει αυτές τις ε, διαπραγματεύσεις. Οπότε νομίζω ότι διασφαλίζονται τα όσα είπαν οι συνάδελφοι και χαίρομαι για το ότι το θέμα αυτό θα περάσει από την Επιτροπή μας χωρίς τριβές. Σας ευχαριστώ. Προθεσμία για τροπολογίες είναι στις 18 Νοεμβρίου 5 ώρα το απόγευμα. Η εξέτασή του θα γίνει στις 20 Ιανουαρίου, ψηφοφορία στην Επιτροπή 21 Ιανουαρίου. Εντάξει. Ωραία. Συνεχίζουμε. Ευχαριστούμε κύριε Φέρμπερ. Με συγχωρείτε. Nous passons aux Personne n'a entendu, Περνάμε στα αποτελέσματα της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του μηχανισμού δυσυνέντας στην Ευρώπη του 2019. Θα εξετάσουμε πολύ προσεκτικά τα σχέδια τα οποία επέλεξε η Κομισιόν για να συγχρηματοδοτηθούν και έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας σήμερα εκπροσώπηση Κομισιόν τον κύριο Ολιβιέ Σιλά συγκεκριμένα. Πού είστε? Ακόμα καλύτερα. Και τον κύριο Χέραν Λότο, παρακαλώ πολύ, ελάτε να εδώ να μας κάνετε την παρουσίαση. Monsieur Ralrotter, je vais vous demander de bien vouloir nous faire cette présentation. Δέκα λεπτά σας δίνουμε για να κάνετε την παρουσίαση. Για να συζητήσουμε μετά και όλα αυτά τα σχέδια. Έχετε το λόγο. Euh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που μου δίνετε να σας παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα αυτής της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων 2019 και αν μου επιτρέπετε θα κάνω την παρουσίαση στα αγγλικά μια και τα, η διαφάνιση είναι στα αγγλικά. Ε, Κυρίε και κύριοι, για να σας ε, παρουσιάσω το αποτέλεσμα της ε, πρόσκλησης αυτής θα ήθελα της προκήρυξης ε, να σας παρουσιάσω εν το τι έχει γίνει στο πρόγραμμα συνδέοντας την Ευρώπη το που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή και μετά να έρθουμε στα αποτελέσματα. Όπως βλέπετε στη διαφάνεια αυτή, η διάδρομη για τα διευρωπαϊκά δίκτυα και το βασικό δίκτυο είναι ένας τομέας κλειδί. Κυρίως εστιάζουμε στις διασυνοριακές διασυνδέσεις, τους χαμένους κρίκους και τις στενοπούς και έχουμε βεβαίως και τις οριζόντιες προτεραιότητες Δηλαδή διαλειτουργικότητα, εναλλακτικά καύσιμα, RTMS SSR κτλ. Και εστιάζουμε ιδιαίτερως στους ε, βιώσιμους τρόπους μεταφοράς όπως βλέπετε και από τις εικόνες. Μάλιστα, αυτό γίνεται μέσω δύο μέσων ε, των πολιετών προκηρύξεων που αφορούν ακριβώς ε, τους διαδρόμους και τις οριζόντιες προτεραιότητες. Ενδεικτικός προπολογισμό είναι στο 95%, αυτή τη στιγμή στο 97% στόχο και βεβαίω έχουμε και τι ετήσιες ε, προκηρύξεις για το συνολικό δίκτυο για τις πιο μικρές διασυνδέσεις ε, και εκεί πέρα ασχολούμαστε με έργα μικρότερη κλίμακα ε, maximum τριών ετών και ο ενδεικτικός στόχος του 5% που είχαμε θέσει είναι στο 3% αυτή τη στιγμή. Εάν δούμε λοιπόν το που βρισκόμαστε στην εφαρμογή του σχεδίου συνδέοντας την Ευρώπη, βλέπετε στις διαφορετικούς αριθμούς από το 2014 στην αρχή όταν ξεκίνησε μέχρι το που βρισκόμαστε τώρα. Ο συνολικός φάκελος ήταν 30 δισεκατομμύρια και βλέπουμε εκεί πέρα ότι μοιράζεται σε μεταφορές, ενέργεια και ψηφιακά. Οι μεταφορές είχαν 23 δισεκατομμύρια και Υπάρχει ένα κομμάτι γενικό και ένα κομμάτι συνοχής. Αυτό έχει ήδη κατανεμηθεί σε προγράμματα εργασίας. Βλέπετε όμως ότι δεν έχουν όλα πληρωθεί ή δεσμευτεί ακόμα. Οπότε ακόμα και αν ε, είχαμε αυτή τη στιγμή υπογράψει 750 συμφωνίες για επιχορηγήσεις, δεν έχουν ακόμα όλα εκταμιευθεί από πλευράς μας, κάτι το οποίο μας επιτρέπει να εφαρμόσουμε την αρχή του «εάν δεν τα χρησιμοποιείς, τα χάνεις». Και θα επανέλθω σε αυτό το τέλος παρουσίασής μου. Εάν ε, δείτε μετά το πώς κατανέμεται στους διάφορους τομείς προτεραιότητας, βλέπετε σαφώς, όπως είπα, ότι τα περισσότερα πηγαίνουν σε μέσα μεταφοράς φιλικά προς το περιβάλλον. Βλέπετε να κυριαρχεί ο σιδηρόδρομος, οπότε από τα 700, τις 751 δράσεις, ε, πολλά από τα κονδύλια, πάνω από 15 δισεκατομμύρια πηγαίνουν στους σιδηροδρόμους ε, και η συνολική αυτή χρηματοδότηση από όλες τις πλευρές, ε, τα 22,3 δισεκατομμύρια που υπάρχουν, έχουν καταλήξει σε 47 δισεκατομμύρια συνολικές επενδύσεις και βεβαίως η βιώσιμη, τα βιώσιμα μέσα μεταφοράς είναι γύρω στο 70% αυτών. Οπότε αυτή είναι η γενική εικόνα και περνάμε τώρα στα αποτελέσματα της προκήρυξης του 2019. Προθεσμία ήταν στις 24 Απριλίου, προϋπολογισμός 100 εκατομμύρια και είχε δύο τομείς προτεραιότητας. Ο ένας ήταν το διασυνοριακό κομμάτι και το άλλο, αυτό εκεί πέρα περιλαμβάνονται και τα λιμάνια και το άλλο αφορά την μείωση του θορύβου από τις εμπορικές αμαξοστοιχίες με 65 και 35 εκατομμύρια αντιστοίχως προπολογισμό. Το βλέπετε αυτό εδώ πέρα. Μιλάμε για ετήσιο διαγωνισμό για το συνολικό δίκτυο. Εάν δούμε μετά τα αποτελέσματα των διαφόρων προτεραιοτήτων, βλέπετε στη διαφάνεια 35 εκατομμύρια για τον θόρυβο των σιδηροδρόμων δεν έχουν ακόμα διανεμηθεί πλήρως γιατί επιλέξαμε προτάσεις για το ποσό των 19 εκατομμυρίων οπότε έχουμε εδώ πέρα μια διαφορά 15 εκατομμυρίων μεταξύ ενδεικτικού και πραγματικού προπολογισμού. Αλλά βεβαίως όταν μιλάμε για το δίκτυο το οποίο περιλαμβάνει διασυνδέσει και λιμάνια είχαμε πολύ μεγαλύτερες ε, προσφορές, ε, κατά 32 εκατομμύρια δηλαδή. Κάτι το οποίο μας δίνει το συνολικό αποτέλεσμα. 39 έργα έχουν επιλογή με συνολικό ύψο 117 εκατομμύρια. Αυτό γίνεται χάρη στο κείμενο της προκήρυξης, μας επιτρέπει μια ευελιξία 20% και αν έχουμε υψηλή προσθέμενη κοινοτική αξία τα διατηρούμε. Ε, μας δίνει την δυνατότητα δηλαδή αυτή το πρόγραμμα. Να σας δώσω τώρα κάποια παραδείγματα έργων που έχουν επιλεγεί. Το πρώτο είναι στον τομέα προτεραιότητα για τον θόρυβο των εμπορικών αμαξιοστοιχείων. Βλέπετε αρκετά κράτη-μέλη από την Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ιρλανδία, Ιταλία και Λουξεμβούργο, Σλοβακία. Καλύπτεται λοιπόν εδώ πέρα ο εξυγχρονισμός του τροχαίου υλικού με διαφορετικά φρένα, υλικά τριβής και νομίζω ότι έχουμε καλύψει τώρα τον τομέα προτεραιότητας αυτών. Μετά έχουμε τον δεύτερο τομέα προτεραιότητας, να σας δώσω και εδώ κάποια παραδείγματα έργων. Το πρώτο έχουμε ένα διασυνοριακό έργο μεταξύ Βρέμης και Χρόνιγκεν, Γερμανίας και Ολλανδίας, με μια στήριξη 12 εκατομμυρίων για μια συνολική επένδυση, ε, επένδυση και το επόμενο είναι πάλι σιδηροδρομικό έργο. Εδώ είναι μια μελέτη όμως μεταξύ Αυστρίας και Ουγγαρίας. Μελέτη η οποία θα γίνει την επόμενη περίοδο για 3,25 εκατομμύρια ευρώ. Συνολική επένδυση 6,5 εκατομμύρια και προετοιμάζεται έτσι το έδαφος για την επόμενη περίοδο για να περάσουμε σε έργο. Μετά, να σας δείξω εδώ ένα έργο σε λιμάνι το λιμάνι του Ούλου στη Βόρεια Φιλανδία όπου γίνονται έργα υποδομών για να αυξηθεί η πρόσβαση και η αποτελεσματικότητα του τελευταίου χιλιόμετρου σιδηροδρομικών διασυνδέσεων. Μια επένδυση 2 εκατομμυρίων και από το ΣΕΦ και 10 εκατομμυρίων συνολικά. Και το τελευταίο έργο που θα σας δείξω εδώ είναι το λιμάνι της ε, Τσιβιταβέκια όπου επίσης ε, έχουμε στήριξη ε, για την αναβάθμιση των σιδηροδρομικών διασυνδέσεων γιατί αυτό το τελευταίο κομμάτι συνήθως δεν λειτουργεί. Και τέλος, κυρία Πρόεδρε, έχω δύο ακόμα διαφάνειες, τρεις, για το τι θα γίνει στο μέλλον για να ενημερώσουμε τους βουλευτές για το τι θα γίνει στο τελευταίο 1,5 έτος του τρέχοντος ε, ΠΔΠ. Όπως είπα στην αρχή υπάρχει πάντα αυτή η αρχή του όποιος δεν τα χρησιμοποιεί τα χάνει τα λεφτά και έχουμε έργα τα οποία δεν εκταμιεύουν τα χρήματα εγκαίρως και καθώς η υπηρεσία μας παρακολουθεί προσεκτικά όλα και τα 751 έργα εξετάζονται όλα και συμφωνούμε μετά με τους δικαιούχους ότι αν δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα κονδύλια επανέρχονται. Έχουμε λοιπόν εδώ πέρα 1,4 εκατομμύρια, μια προκήρυξη που συμφωνήσαμε τα κράτη-μέλη και έγινε στις 16 Οκτωβρίου με προθεσμία υποβολής προσφορών στις 26 Φεβρουαρίου. Και εδώ πέρα βλέπετε πρώτα απ' όλα Έχουμε έργα στους διαδρόμους του βασικού δικτύου, η προτεραιότητα η οποία δεν είχε ανοίξει από το 2014, η πρώτη προκήρυξη για τον γενικό φάκελο και από το 2015 για τον φάκελο της συνοχής. Και άρα υπήρχε αίτημα αν ε, έστρεφαν λεφτά να ξαναπέσουν εδώ και βλέπετε προτεραιότητες επίσης για πρωτότυπα RTMS για ασφαλείς υποδομές, ε, κυρίως ε, πάρκινγκ ε, και διάφορες δραστηριότητες στον τομέα της λειτουργικότητας ITS και ΣΕΖΑΡ και βέβαια αυτό το οποίο βλέπουμε εδώ είναι η αστική κόμβη και η λεωφόρη της θάλασσας. Αυτά νομίζω καλύπτουν επαρκώς την ε, περίοδο που απομένει στο τρέχον ΠΔΠ και θα προετοιμάσουμε την επόμενη περίοδο. Και τελευταία διαφάνεια αφορά ακριβώς ε, την ε, εγκατάσταση αυτή, την διευκόλυνση όπου έχουμε χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, το Ταμείο Στατικών Επενδύσεων πιθανώς, και αυτό μπορεί να γίνει είτε μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων είτε των Εθνικών Τραπεζών ή και του ιδιωτικού τομέα. Έχουμε λοιπόν 200 εκατομμύρια το ERTMS και τα εναλλακτικά καύσιμα. Αναμένουμε η προκήρυξη να γίνει το Νοέμβριο, πιθανώς στις 15, αλλιώς 1η Δεκεμβρίου Έχουμε λοιπόν έναν διαφορετικό τρόπο εργασίας ε, γιατί θα έχουμε ένα πρόγραμμα τριμηνιαίο και τρέχον για να αντιμετωπίσουμε συγκεκριμένες προτεραιότητες ε, στο όλο που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν μέσω των κανονικών προκηρύξεων του ΣΕΦ. Ένα συμπληρωματικό εργαλείο και το αντιμετωπίζουμε που σας είπα με αυτήν την εγκατάσταση. Σας ευχαριστώ λοιπόν για το χρόνο που μου δώσατε για να σας εκθέσω τις εξελίξεις ε, στο τρέχον τη ΔΕΛΤΑΠΗ και το τι γίνεται στο 2019. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ξεκινάμε τη συζήτηση αμέσως. Κύριε Μαρινέσκο, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ για αυτή την παρουσίαση. ποιο είναι το επίπεδο των ποσών που θα ανακτήσετε από σχέδια τα οποία δεν εφαρμόζονται, δεν υλοποιούνται, στο άμεσο μέλλον. Ποιες είναι οι χώρες οι οποίες κινδυνεύουν να μην χρηματοδοτηθούν. Αν υπάρχει διαφορά ανάμεσα στα ταμεία συνοχής και, την, και το μηχανισμό και τα ποσά του μηχανισμού σύνδοδος στην Ευρώπη. Μετά, σε αυτή την ε, πρόσκληση υποβλήθηκαν πολλές μελέτες. Μελέτες οι οποίες θα υλοποιηθούν πότε. Γνωρίζετε ότι κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για το ε, ΣΕΦ 2 το συζητήσαμε. Είχαμε πει ότι το Κοινοβούλιο θέλει μελέτες οι οποίες θα υλοποιηθούν όμως σύντομα. Όχι μελέτες γενικώ και αορίστως για το μέλλον. Μόνο για να πάρουν τα λεφτά. Merci Πρόεδρος, ευχαριστώ κύριε Μαρινέσκο. Κύριε Ντάνιελσον, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ και εγώ για την παρουσίαση. θα έκανε και εγώ την ίδια ερώτηση με τον κύριο Μαρινέσκο. Ποιε είναι οι χώρε οι οποίε κινδυνεύουν να χάσουν τα χρήματα, τη χρηματοδότησή του, λόγω μη υλοποίηση. Επίση, θα ήθελα να ρωτήσω, ποιοι είναι οι βασικοί λόγοι κατά την άποψη τη Κομισιόν που χώρε, κάποιε χώρε, υποχρησιμοποιούν τα ποσά τα οποία του έχουν καταλογιστεί. και είναι πολύ καλό που προσπαθούμε του χρόνου να δώσουμε μεγαλύτερα κονδύλια για το βασικό δίκτυο. Ο κ. Δίας. Θα μιλήσω ισπανικά. Καταρχήν να ευχαριστήσω την Κομισιόν για την παρουσίαση αυτή. Πέραν, ε, αντί για ερωτήσεις, θα ήθελα να εκφράσω την εξή σκέψη. Προκειμένου να καταλάβει η Κομισιόν πόσο σημαντικό είναι να βελτιωθούν μερικές συνδέσεις. Και άλλοι συνάδελφοι, είχαμε πάει την περασμένη εβδομάδα στις χώρες μας, στις εκλογικές μας περιφέρειες κλπ. Και την προηγούμενη εβδομάδα επισκέφθηκα την Εξτρεμαδούρα, μια από τις πιο απομονωμένες περιοχές της Ευρώπης. Η ε, πρωτεύουσα είναι η Μέριδα, την επισκέφθηκα από την ρωμαϊκή εποχή ονομαζόταν Εμέριτα Αουγούστα. Ήταν από τις πόλεις, τις πιο καλά συνδεδεμένες πόλεις της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, με τη Ρώμη και με άλλα μέρη της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, πριν από 2.000 χρόνια βέβαια. Αυτή τη στιγμή τα πράγματα είναι ακριβώς αντίθετα. Η Εστρεμαδούρα είναι πλέον περιβόητη στην Ισπανία και στην Ευρώπη ως μία από τις πιο απομονωμένες σιδηροδρομικά περιοχές της Ευρώπης και όχι μόνο από την, Ισπανία, από την υπόλοιπη Ισπανία, αλλά και από την διπλανή της Πορτογαλία. Ε, τα τρένα ε, στην Στρεμαδούρα αποκαλούνται τρένα της ντροπή, ε, γιατί είναι λίγα τα δρομολόγια, καθυστερημένα, πολύ συχνά γίνονται, παρουσιάζονται βλάβες, επεισόδια, Κάτι που δημιουργεί σημαντικό πρόβλημα προφανώς. Θα ήθελα λοιπόν να εκφράσω εδώ τη φωνή των ανθρώπων από την Εστρεμαδούρα και ενδεχομένως και από την Πορτογαλία. Θα πρέπει η Κομισιόν να αντιληφθεί την ανάγκη να βελτιωθούν αυτά τα δρομολόγια, γιατί αυτά τα δρομολόγια βοηθούν όχι μόνο μία χώρα, αλλά δύο, και την Ισπανία και την Πορτογαλία. Και όχι μόνο αυτές τις δύο, διότι συνδέουν όλο τον Νότο με την υπόλοιπη Ευρώπη. Οπότε δεν έχω ερωτήσεις να σας κάνω, απλά προσπαθώ να σας ευαισθητοποιήσω στην παρουσίαση μελλοντικών σχεδίων. Ε, δεν χρειάζεται απλώς να βελτιώσουμε την ποιότητα. Θα πρέπει να συνεχίσουμε αυτό που ξεκίνησαν οι Ρωμαίοι 2.000 χρόνια πριν και αυτή τη στιγμή ε, βρίσκεται σε μια κατάσταση στάσιμη εδώ και πολύ καιρό. Ευχαριστώ πολύ και συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δίας και κυρία. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Δεν θέλω να ευχαριστήσω την Επιτροπή για αυτή την αναλυτική παρουσίαση. Χρήσιμο να έχει κανείς διαφάνειες που συνοπτικά και ξεκάθαρα να παρουσιάζουν τα διάφορα ζητήματα. Η βασική μου ερώτηση είναι η εξής. Πώς θα πρέπει να εξελιχθεί η διευκόλυνση συνδέοντας την Ευρώπη, για να εξυπηρετήσει αυτή τη νέα συμφωνία που έχουμε, ότι μέχρι το 2050 θα πρέπει να έχουμε ε, πάψει να βασιζόμαστε στον άνθρακα. Έχουμε πολλές συζητήσεις και πολλές φορές έχουμε ακούσει για τις ε, χρηματοδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, η οποία πηγαίνει μόνο προς project τα οποία είναι οδέτερα προς τον άνθρακα. Όμως, σε ορισμένες περιπτώσεις αυτά τα έργα ε, είναι έργα που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ανάπτυξη του οδικού δικτύου. Βλέπετε λοιπόν να έχει μεταβληθεί ή να πρέπει να μεταβληθεί με κάποιον τρόπο η πολιτική της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων στο θέμα αυτό. Ένα άλλο ζήτημα που ήθελα να θίξω είναι το θέμα του θορύβου. Μιλήσατε για τη χρηματοδότηση, για την προστασία, την αντιμετώπιση του θορύβου. Ε, φαντάζομαι ότι σε ολόκληρη την Ευρώπη υπάρχει όλο και μεγαλύτερη ανησυχία για την ρήπανση από θόρυβο, ιδιαίτερα στις αισθητικές περιοχές. Έχουμε όλο και περισσότερες επιστημονικές μελέτες που δείχνουν ότι έχει αντίκτυπο ο θόρυβος στην ανθρώπινη υγεία. Θα ήθελα να με ενημερώσετε αν έχει υπάρξει ε, και αν γίνονται μελέτες για τον θόρυβο που θα προκαλέσουν τα διάφορα έργα που χρηματοδοτούνται. Κύριε Ζήλη, το ECR, ε ευχαριστώ. Το τον εκπρόσωπο της Επιτροπής για αυτή την πολύ ε, πλήρη παρουσίαση. Η ερώτηση δική μου είναι παρόμοια με εκείνα του κυρίου Μαρινέσκου. Δεν με ενδιαφέρει ιδιαίτερα να ακούσω ποιε χώρε είναι αυτέ που αφορά το πρόβλημα, αλλά μιλήσατε για ότι το 61% είναι ποσά τα οποία έχουν δεσμευτεί και, ότι και οι πληρωμές είναι στο ύψος του 31%. Θα ήθελα όμως να μου πείτε τι προβλέπετε για την ολοκλήρωση αυτού του PDP. Αν μπορείτε να μου δώσετε δηλαδή αυτά τα αντίστοιχα ποσοστά πληρωμών και τουλάχιστον δεσμευμένων ποσών μέχρι το τέλος της, ε, του πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου που προβλέπετε να κυμανθούν. Ε, γιατί αυτό έχει μεγάλη σημασία όταν προετοιμάζουμε και το νέο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, δηλαδή από την εμπειρία που αποκτήσατε από το τρέχον δημοσιονομικό πλαίσιο. Έχετε εντοπίσει κάποια συγκεκριμένα προβλήματα που να οδηγούν στην μη απορρόφηση των κονδυλίων. έτσι ώστε να φροντίσουμε να, αντιμετωπιστούν αυτά για το ΣΕΦ την επόμενη χρονιά. Η κυρία Κουντουρά. Να ευχαριστήσω την Κομισιόν για την παρουσίαση αυτή και θα ήθελα να τοποθετηθώ και να κάνω και μία ερώτηση. Η συντριπτική πλειοψηφία των έργων που προτείνονται για χρηματοδότηση παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον, ενώ είναι σαφής ο προσανατολισμός τους προς περισσότερες σιδηροδρομικές μεταφορές. Κάποια έργα μάλιστα παρουσιάζουν και γεωστρατηγικό ενδιαφέρον, όπως είναι η σιδηροδρομική σύνδεση Πυθίου Ορμενίου στην βορειοανατολική Ελλάδα. Οι ανάγκες όμως είναι τεράστιες και παρά τα όποια βήματα γίνονται, είμαστε ακόμα μακριά από το να πετύχουμε βιώσιμες μεταφορές στην Ευρώπη τη στιγμή που η κλιματική κρίση θα εντείνεται. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω αν εκτιμάτε ότι είναι εφικτό να πετύχουμε τους στόχους μας για το κεντρικό και το εκτεκταμένο δίκτυο με τους σημερινούς ρυθμούς ολοκλήρωσης και αν εκτιμάτε ότι οι τεχνολογικές καινοτομίες τα επόμενα χρόνια, όπως μεγαλύτερη διείσδυση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις μεταφορές, θα μας αναγκάσουν να αναθεωρήσουμε τις προτεραιότητές μας αναφορικά στα δίκτυα υποδομών, που θα μας επιτρέψουν να πετύχουμε ένα σύστημα μεταφορών με μηδενικές εκπομπές ρήπων μέχρι το 2050. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Ρικέ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ και τον εκπρόσωπο της Επιτροπής για την παρουσίαση. Ήταν πολύ διαφωτιστική. Έχω τρία ερωτήματα. Πρώτον, τι θα γίνει με αυτή τη ε, μεταφορά κοντιλίων στην οποία αναφερθήκατε. Δηλαδή, ε, υπάρχει ένα συγκεκριμένο έργο από το οποίο, ε, στο οποίο διαπιστώνουμε ότι μπορούν να κρατηθούν χρήματα και αυτό γίνεται δηλαδή αναέργο ή στο σύνολο του προϋπολογισμού. με λίγα λόγια, αυτέ τι μεταφορέ δηλαδή χρημάτων που δεν απορροφήθηκαν, τι ελέγχετε και τι φροντίζετε να γίνουν ανά project ή συνολικά. Δεύτερο ερώτημα. Έχει σχέση και με την τελευταία σας διαφάνεια. Η διευκόλυνση για την συγχρηματοδότηση, το blending facility. Αυτό είναι ένας μηχανισμός που επιτρέπει μια χρηματοδότηση κατά τη διάρκεια του 2019. Θα ήθελα να μου πείτε αν αυτό το ποσό έχει ε, ε, υπολογιστεί με τρόπο που να βασίζεται σε μια αξιολόγηση των αναγκών και αν αυτό που διαπιστώσαμε το 2019 θα το δούμε και στις επόμενες χρονιές. Τρίτο ερώτημα διαπιστώνω ότι είναι λίγα τα έργα που χρηματοδοτούνται για την αντιμετώπιση του θορύβου από τις σιδηροδρομικές μεταφορές. Παρά το γεγονός ότι είχαν γίνει πολλές επενδύσεις ε, ε, δισεκατομμυρίων. Και θυμίζω ότι υπήρχαν κράτη-μέλη όπως η Γερμανία που είχαν επισημάνει πόσο σημαντικό είναι να δώσουμε τέτοιες χρηματοδοτήσεις και πόσο σημαντικό είναι το θέμα. Πώς γίνεται λοιπόν ένα ζήτημα να έχει αναδειχθεί ω τόσο σημαντικό και να μην είχαν υπάρξει προτάσεις για έργα τα οποία να το αντιμετωπίζουν. Ευχαριστώ κύριε Ρικέ. Και εγώ θέλω να μιλήσω, γιατί είναι σημαντικό το θέμα. Σήμερα ε, ζούμε μια εποχή, ένα συγκεκριμένο μήνα. Ε, ο Οκτώβριος ήταν ο πιο ε, ζεστός μήνας, πιο ζεστός Οκτώβριος ε, στην ιστορία της Ευρώπης. Συν το ότι έχουμε τις φυσικές καταστροφές, τις θεομηνίες, πλημμύρες, ξηρασίες, φωτιές. Οι οδικές μεταφορές έχουν τρομακτική επίδραση στο περιβάλλον, 30% των εκπομπών του διοξιδίου του άνθρακα ε, και το σχέδιο είναι να φτάσουμε στην μηδενική εκπομπή. Έχει γίνει προσπάθεια. Έχει γίνει προσπάθεια, είναι αλήθεια. Έχουμε επενδύσει περισσότερο στις ε, σιδηροδρομικές μεταφορές, αλλά το πρόβλημα είναι οι οδικές μεταφορές και εκεί είναι το νούμερο δύο στις επενδύσεις μας. Πού πραγματικά είναι οι πραγματικές αναλυτικές λύσεις. Υπάρχουν, αλλά, είναι, αλλά χρηματοδοτούνται με πολύ μικρότερα ποσά οι εσωτερικές πλωτές οδοί, ας πούμε. Το θαλάσσιο και οι πλωτές οδοί είναι ένα πολύ μικρό ποσοστό. Εδώ θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας, να κάνουμε πρόοδο εκεί πέρα. Να... Δεύτερον, στην παρουσίασή σας δεν αναφέρεται το ζήτημα, πολύ καυτό είναι στην Ευρώπη, η χειροτέρευση των υποδομών στην Ευρώπη. Γυράσκουν οι υποδομές μας και στο σιδηροδρομικό δίκτυο και στο οδικό δίκτυο. Ο μηχανισμός διασύνδεσης Ευρώπης δεν θα έπρεπε να είναι παρόν και εκεί. Δεν τον βρίσκω όμως. Η δεύτερη μου λοιπόν ερώτηση είναι πώς μπορούμε να επενδύσουμε στην κινητικότητα της καθημερινότητας των πολιτών μας. Τι κάνουμε εμείς για το σήμερα, για την κινητικότητα των πολιτών μας σήμερα. Τρίτο θέμα που θέλω να θίξω Νομίζω ότι έχει έρθει η στιγμή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταλάβει ότι οι μεταφορές θα πρέπει να επηρεάζουν το έργο και των υπόλοιπων επιτρόπων και των υπόλοιπων επιτροπών επίσης. Για παράδειγμα, Πράσινη Συμφωνία, Green Deal, πολύ ωραίο, το έχει ανακοινώσει η καινούργια επιτροπή. Πώς όμως η Επιτροπή θα εντάξει μεταφορές εκεί. Για παράδειγμα, εναλλακτικά καύσιμα. Κάνετε κάποια προβολή στο μέλλον για τη χρήση του υδρογόνου. Για να δημιουργηθεί μια ολόκληρη βιομηχανία του υδρογόνου. Αυτά είναι τα πραγματικά οραματικά σχέδια. Στο Green Deal υπάρχει επίσης και όλο το θέμα των νεοτερισμών. είχατε μια διαφάνεια για το ψηφιακό, για το ψηφιακό κομμάτι. Στο ψηφιακό κομμάτι δεν γίνονται πραγματικές επενδύσεις. Αν θέλω δηλαδή εγώ να βγω, να πάρω το τρένο και να, μετά το τρένο να πάρω ένα ποδήλατο ή να μοιραστώ ένα αυτοκίνητο κλπ. Εκεί θα έπρεπε να μπει το ψηφιακό κομμάτι. Πώς θα προσανατολίσετε λοιπόν αυτές τι επενδύσει έτσι ώστε να απαντήσουμε και τις κλιματολογικές, ε, τα κλιματολογικά προβλήματα και τα ψηφιακά θέματα και ταυτόχρονα να στηρίξουμε και την καθημερινή κινητικότητα των ανθρώπων. Αυτό περιμένω από εμάς. Κύριε Σοντέ, σα έχω σημειώσει, αλλά είστε πιο κάτω στον κατάλογο. Ο κύριο Νάμποκοφ. Thank you very much, Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Εδώ, εδώ είμαι. Πρώτα απ' όλα σας ευχαριστώ κύριε Ράιτερς για την παρουσίαση που κάνατε και πρέπει να πω ότι το μέσο συνδέοντας την Ευρώπη μαζί με το Erasmus Plus είναι ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης γιατί εφαρμόζει έργα τα οποία είναι συμβολικά για τις ε, τοπικές ε, κοινωνίες. Και θα ήθελα να σας πω ότι η οικογένειά μου στο παρελθόν είχαν εργαστεί στους πρώτους σιδηρόδρομους της χώρας μου και ακριβώς στην ίδια διαδρομή τώρα, χάρη σε αυτό το μέσο, θα δούμε τρένα που θα ταξιδεύουν με 200 χιλιόμετρα την ώρα. Ε, Κατ' θα αλλάξει τις ζωές των ανθρώπων που ζουν εκεί. Κυριολεκτικά θα αλλάξει τις ζωές τους περιοχές ε, που ε, τι οποίε έχει εγκαταλείψει ο κόσμο ε, λόγω έλλειψης θέσεων εργασία ή άλλων συνθήκων, μπορούν και πάλι να προσελκύσουν ανθρώπους γιατί είναι γρήγορο και εύκολο να ταξιδέψει κανείς στις μεγάλες πόλεις για να δουλέψει. ακριβώς λόγω των γρήγορων τρένων και το ερώτημά μου αφορά το μέλλον αυτού του μέσου και εδώ πέρα μιλάω ως εισηγητής ε, για το CPR και το μέλλον της πολιτικής συνοχής. Γιατί υπάρχει αυτή η υποχρηματοδότηση και βασίζεται στο να βρει 10 δισεκατομμύρια από το Ταμείο Συνοχής. Εάν είναι τόσο σημαντικό και όλοι συμφωνούμε ότι το πρόγραμμα πρέπει να συμφωνήσει και να εφαρμόζει τόσο σημαντικά έργα τα οποία επηρεάζουν και το περιβάλλον, γιατί γνωρίζουμε ότι οι σιδερόδρομοι είναι πολύ φιλικοί προς το περιβάλλον. Γιατί υπάρχει αυτή η υποχρηματοδότηση εξ αρχής. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Τζέπαρνε, έχει τον λόγο. Ναι, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κύριε Ρόιτρες. Έχω τρεις σύντομες ερωτήσεις. Για ποιους λόγους ε, δεν έχουν προκηρυχθεί τα προγράμματα για τη μείωση του θορύβου των εμπορικών ε, αμαξοστοιχείων. Υπάρχει πρόβλημα ανταγωνισμού, παραδείγματο χάρη. Ε, βλέπουμε, παραδείγματο χάρη στη Γερμανία, πως οι εταιρείε προτιμούν να ασχοληθούν με οδικά έργα και δεν υπάρχει το εργατικό δυναμικό να κάνει τέτοια περίπλοκα σιδηροδρομικά έργα. Ε, επίσης ε, θα πρέπει να κλείσουν ακριβώς αυτά τα κενά, τα διασυνοριακά βασιζόμενοι στην εμπειρία που έχουμε. Και τρίτη ερώτηση, τι γίνεται με τον εξηλεκτρισμό του σιδηροδρομικού δικτύου. Εκεί πέρα ως πράσινοι θεωρούμε ότι υπάρχουν πάρα πολλές δυνατότητες για μείωση των εκπομπών και για να περάσουμε στην ε, κινητικότητα στον τομέα των σιδηροδρόμων. Σας ευχαριστώ κυρία Τεπαρνέ. Κυρία Γκαρσία Μινιός, έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ πολύ την Κομισιόν για την παρουσίαση και για το γεγονός ότι έχει δει τη σημασία του Κανφραν ε, στην ε, διασυνοριακή σύνδεση Ισπανίας και Γαλλίας και την ανάγκη να βελτιωθεί η διοικητική συνεργασία σε τέτοιου είδους ε, σχέδια κοινού ενδιαφέροντος. Όπως είπε ο κ. Μπάουθα προηγουμένως, για την ε, έλλειψη σύνδεση μεταξύ συγκεκριμένων περιοχών. Να υποφεληθώ και εγώ για να τονίσω τη σημασία ε, τη, του διαδρόμου Κανταβρίας Μεσογείου. Ε, η επαρχία του Τερουέλ στη Γανία, στη, στην Ισπανία έχει τα ίδια ακριβώ προβλήματα αυτά που είπε ο κύριος, ο συνάλφος, για την Εξτρεμαδούρα. Κυρία Ντεσόντε, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Μιλήσατε για την κινητικότητα και πολύ σωστά μιλήσατε ε, για τις διάφορες καταστροφές που έχουν γίνει μεταξύ αυτών και τις γέφυρες της ε, ε, της Γένοβας. θα ήθελα να σας δώσω ένα πολύ συγκεκριμένο παράδειγμα. Στο Φρέζους είναι, έχουμε μια γέφυρα για οχήματα, ποδήλατα και πεζούς. Είναι η γέφυρα de la ε, βρίσκεται σε πολύ κακή κατάσταση. Πρέπει να επανακατασκευαστεί επιγόντως. Εδώ όμως και 10 χρόνια αδυνατούμε να προχωρήσουμε. Γιατί, Γιατί ε, η γέφυρα βρίσκεται σε μια περιοχή προστασίας του περιβάλλοντος, προστασίας των, της ε, πανίδας και άλλων σημαντικών πραγμάτων τα οποία πρέπει να προστατευτούν. Όμως είναι απολύτως απαραίτητο να ληφθεί υπόψη η ασφάλεια των ανθρώπων. Πρέπει να μας βοηθήσετε εσείς από την Κομισιόν να προχωρήσουμε ε, πέραν της προστασίας μερικών φιδιών. Προσοχή με τα φίδια λέει η Πρόεδρος, είναι απόλυτος απαραίτητα για τους βιοτόπους μας. Χωρίς την βιοπικιλότητα δεν μπορεί να ζήσει ο άνθρωπος. Ναι, αλλά οι άνθρωποι χρειάζονται ταυτόχρονα και να μπορούν να περάσουν και τη γέφυρα. Κομισιόν, πολλές ερωτήσεις, λίγος ο χρόνος, λυπάμαι. Δύο θέματα επανέρχονται. Οπότε να ξεκινήσω με αυτά με περισσότερες λεπτομέρειες. Ο κ. Μαρινέσκου λέει ποιο ποσό εκτελείται ο προπολογισμό μας και πώς ε, ε, ανακτούμε ποσά, πόσα ποσά, ε, ποιες χώρες και η διαφορά μεταξύ γενικού προπολογισμού και προπολογισμού συνοχής. από την παρουσίασή μου αντιλαμβάνεστε ότι η πρόσκληση που έγινε είναι ισορροπημένη μεταξύ των μεταξύ του γενικού προπολισμού και του προπολισμού συνοχής. Δεν είναι δηλαδή αλήθεια ότι οι χώρε συνοχής ε, τα πάνε καλύτερα ή χειρότερα. Όλες οι χώρες βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο, αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα στην υλοποίηση των σχεδίων. Τα βασικά προβλήματα που οδηγούν σε καθυστερήσεις είναι ε, είτε θέματα αδειών, είτε θέματα ε, προμηθειών. Για παράδειγμα, περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις καθυστερούν πολύ, καθώς επίσης καθυστερούν και πολλοί διαγωνισμοί ε, οι οποίοι προσβάλλονται στα δικαστήρια. Η προσέγγιση δική μας δεν είναι να δούμε συνολικά τα ποσά, αλλά ανά σχέδιο. Το κάθε σχέδιο αξιολογείται από μόνο του. Αν δούμε μαζί με το δικαιούχο ότι τα ποσά, τα κονδύλια δεν μπορούν να καταναλωθούν έγκαιρα, τότε τα χρήματα αυτά επιστρέφουν στον προπολογισμό και αυτό γίνεται συνενετικά. Γιατί θα πρέπει να τροποποιηθεί η συμφωνία ε, χρηματοδοτικής βοήθειας, οπότε σε αυτές τις περιπτώσεις συμφωνούν και οι δικαιούχοι. Μόνο με αυτόν τον τρόπο επιστρέφονται τα χρήματα και μετά ξαναβγαίνουν από τον προπολογισμό. Πώς διαφέρει αυτή η φορά από την προηγούμενη. Την προηγούμενη φορά ο προπολογισμό ήταν 8 δι με 20% περίπου ε, ανακτηθέντα ποσά. Τώρα είμαστε 1,4, στο 1,4 δις. Είναι μικρό σχετικά με τον διατεθέμενο προπολογισμό. Και πάλι μπορεί να έχουμε κάποιες επιστροφές στον προπολογισμό, αλλά θα είναι λιγότερε από την προηγούμενη φορά. Ίσως στο μισό αυτού που είχαμε την περασμένη φορά, ίσως δηλαδή γύρω στο 10%, ίσως ούτε καν 10% του προπολογισμού των 1,4 δισεκατομμυρίων. Άρα πάμε καλύτερα. Λογικό, γιατί έχουν οριμάσει πολύ περισσότερα σχέδια, τα κράτη-μέλη έχουν περισσότερη εμπειρία, ακόμα και στι χώρε συνοχή. Αν υπάρχουν μερικέ χώρε που τα πάνε καλύτερα από άλλε, όχι. Όλε οι χώρε έχουν σχέδια με καθυστερήσει. Δεν μπορούμε να πούμε ότι κάποιες χώρες είναι καλύτερες από κάποιες άλλες. Όλες οι χώρε έχουν περίπου την ίδια επίδοση. Δεν μπορώ να σας πω δηλαδή ότι μια χώρα τα πάει πραγματικά πολύ άσχημα ή κάποια άλλη ότι διαπρέπει. Τα κονδύλια θα πρέπει να κατανοηθούν έγκαιρα. Μιλήσατε για τις μελέτες. Ναι, οι μελέτες ε, πρέπει να έχουν υλοποιηθεί μέχρι το 2023, τρία χρόνια μετά δηλαδή. Ακόμα και αυτές που σας παρουσίασα σήμερα, ε, μπορείτε να βρείτε και μια προσούρα ε, στην είσοδο. Η επιλογή είναι πάρα πολύ αυστηρή για τις μελέτες και η οριμότητα των σχεδίων ελέγχεται πάρα πολύ αυστηρά Οι μελέτε θα πρέπει έγκαιρα να ολοκληρωθούν και να οδηγήσουν και σε ολοκλήρωση του σχεδίου μέχρι το 2022 ή 2023. Δηλαδή οι μελέτες μέχρι το 2022-2023 και μετά θα πρέπει και τα σχέδια να ελοποιηθούν ταχύτατα. Δεύτερο σημείο, ο τρόπος που χρησιμοποιούμε τον προπολογισμό και πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την ε, κλιματική συνιστόσα. Να υπογραμμίσω καταρχήν ότι ο εν λόγω προπολογισμό, μιλάμε για ένα, για μία πρόσκληση, άρα σας, αλλά σα έδειξα και τα συνολικά στοιχεία, πάνω από 70%, 71% συγκεκριμένα, ε, στηρίζουν βιώσιμου τρόπους μεταφοράς. Αν δείτε στο θέμα των οδικών μεταφορών, συμφωνώ είναι αρκετά ψηλά τα ποσά, αλλά συμπεριλαμβάνει το ITS, τα, τους χώρους στάθμευσης, ε, την οδική ασφάλεια. Όλα αυτά βρίσκονται στη συγκεκριμένη, στο συγκεκριμένο κονδύλι. Αυτά που είναι πραγματικά και αποκλειστικά υποδομές μεταφορών είναι πολύ λίγα και αφορούν τις ε, χώρες συνοχής σε διαμεθοριακά σχέδια, τίποτα άλλο. Αυτή είναι η προσέγγιση μας. Ε, στο, στην επόμενη περίοδο οι μεταφορές θα βρεθούν στο 75% Οπότε είναι πολύ ψηλό, ελπίζω να το καταλαβαίνετε. Μόνο το ίτερ είναι στο 100%. Η, μετά το ίτερ είναι ο μηχανισμός συνδέοντας την Ευρώπη στο 75%. Ε, Ε, το όλο, ο μηχανισμός θα είναι στο 60%, άρα οι μεταφορές θα πρέπει να είναι στο 75%. Ε, 75% ε, δηλαδή των ποσών να ε, προορίζονται για την κλιματική αλλαγή. στο ψηφιακό κομμάτι την άλλη μεριά ήδη έχετε και τα εναλλακτικά κάψιμα, στις υποδομές τους, και έχουμε μια πολύ καλή επίδοση εκεί πέρα. Κάτι μας οδήγησαν στις διαπραγματεύσεις για το δεύτερο μηχανισμό ασθενότητας στην Ευρώπη, το 85% να πηγαίνουν σε υποδομές και 15% στις υπόλοιπες συνιστώσεις. Αποφασίσαμε στις διαπραγματεύσεις ότι θέλουμε να αυξήσουμε στο 40% το 15%. Σχεδόν τριπλασιασμό δηλαδή αυτού του κομματιού από 85-15 να πάμε σε 60-40. Αυτό ως απάντηση στις ανάγκες ηλεκτροδότησης ε, και στους αυτοκινητοδρόμους αλλά και στον σιδηρόδρομο και να ε, εξασφαλίσουμε ότι θα καλύψουμε και άλλα εναλλακτικά καύσιμα όπως το υδρογόνο. Μετά κάποια πιο συγκεκριμένα σχόλια που έγιναν. Κύριε Μπάουθα και η κυρία Μουνιώθ μίλησαν για τις διασυνοριακές ε, συνδέσεις. Σήμερα σας μίλησα μόνο για αυτή τη συγκεκριμένη πρόσκληση, αλλά η Μέριδα βρίσκονται στον Ατλαντικό διάδρομο και η σύνδεση μεταξύ Εύωρα και Μέριδα, Εύωρα στην Πορτογαλία, Μέριδα στην Ισπανία, είναι κλειδί. Και αν ο κ. Μαρινέσκου ρωτήσει τα τι περιμένουμε, ποια ανακατανομή περιμένουμε θα γίνει σύντομα, αυτή είναι μια, αυτό το σχέδιο είναι μία από αυτές. Ε, το, είναι απόλυτα σημαντικό αυτό το, αυτή η σύνδεση είναι απόλυτα σημαντική, δεν αμφισβητείται καθόλου. Δεν ε, μπορούμε ε, να έχουμε την αισθηματούρα να συνδέεται μόνο με αεροπλάνα το πρόγραμμα εργασία, ο συντονισμό είναι, υπάρχουν, τα χρήματα υπάρχουν. Τώρα πρέπει να δούμε την υλοποίηση του σχεδίου και αυτήν παρακολουθούμε. Αν δεν υλοποιηθεί τώρα, θα δούμε με την Ισπανία και την Πορτογαλία μήπω μπορεί να υλοποιηθεί στο επόμενο πολιτέ δημοσιονομικό πρόγραμμα. Και δεν μιλώ μόνο για τη Μέριδα, έτσι. Σχεδόν όλα μας τα προγράμματα, τα σχέδια μας είναι διασυνοριακά και αυτό περιμένουν οι πολίτες. Μετά, τι κάνουμε για τη συντήρηση, για παράδειγμα, των γεφυρών. Ας είμαστε προσεκτικοί. Ή χρηματοδοτούμε έργα που έχουν σχέση με την κλιματική αλλαγή ή θα κάνουμε πιο πολλά για τους δρόμους. Δεν μπορούμε να κάνουμε τα δύο. Αν θέλουμε να αντικαθιστούμε και τις παλιές γέφυρες, τότε θα πρέπει να αυξήσουμε τα ποσά που χορηγούμε για τις υποδομές. Αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει και ταυτόχρονα να αυξήσουμε και τα ποσά για την κλιματική αλλαγή. Τώρα, από την άλλη μεριά, γίνεται έρευνα για το πώς μπορούμε να ε, παρακολουθούμε την κατάσταση των υποδομών. Μπορούμε να κάνουμε τέτοιου τύπου μελέτες και έρευνες. Ναι, Η, αν μπαίναμε στη συντήρηση θα εξαντλούσαμε τον προπολογισμό μας. Γιατί ήδη λέτε ρωτάτε τι μπορούμε να κάνουμε με τόσο λίγο προπολογισμό. Πρέπει να εστιάσουμε. Εστιάζουμε σε διασυνοριακά σχέδια και πολύ συγκεκριμένα στα σχέδια τα οποία έχουν κλιματική διάσταση. Ανακτικά καύσιμα και τέτοια. Οπότε καταλαβαίνω το αίτημα, αλλά θα πρέπει να είμαστε αυστηροί σε αυτό. Μετά, ε, γιατί δεν είχαμε αρκετές προτάσεις για τον θόρυβο στις δρομικές μεταφορές. Ε, είναι η τρίτη φορά που κάνουμε τέτοια πρόσκληση και αντικαθιστούμε ήδη με αυτόν τον τρόπο το 1 τέταρτο των αντίστοιχων υποδομών φρένων δηλαδή ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε μετακινούμαστε πραγματικά αποφασιστικά σε στόλους που θα, κάνουν, θα δημιουργούν λιγότερο, ε, λιγότερη χορύπανση. Ελπίζουμε ότι από μια στιγμή και μετά η αγορά θα κάνει τη δουλειά μας. Ότι θα απενδύσουμε αρχικά και μετά η αγορά θα κάνει τη δουλειά μας. Κύριε Ζήλε, αν θα είμαστε έτοιμοι για το επόμενο πολιτές δημοσιονομικό πρόγραμμα, ναι, πιστεύω, γιατί σε αυτό τον προπολογισμό ήδη μπορούμε να τον εκτελέσουμε καλύτερα από τον προηγούμενο και την επόμενη φορά θα είμαστε ακόμα καλύτεροι γιατί όλα τα σχέδια υπό το τρέχον πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο έχουν κάποιες φορές καθυστερήσεις, αλλά όταν ε, λυθούν τα προβλήματα αδειοδότησης και προμηθειών, όλα αυτά τα σχέδια θα περάσουν στην εκτέλεση. Οπότε κύριε Νόβακοφ, ναι, θα έχουμε σημαντική ανάγκη στήριξης διασυνοριακών σχεδίων. Ε, γιατί η τάση των κυβερνήσεων είναι να ξοδεύουν τα ποσά σε εθνικά σχέδια. Αν δεν είμαστε εμεί εκεί να παρακολουθούμε, δεν θα έχουμε αρκετά διασυνοριακά. Και ήδη μπορώ να σας, ήδη μπορώ να σας πω πόσα θα χρειαστούμε για τέτοιου είδους σχέδια στην επόμενη περίοδο. Νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο κλείνω. Απάντησα πρέπει να έχω απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις, Πρόεδρε. Merci beaucoup. Και εμείς σας ευχαριστούμε για αυτή την συνολική παρουσίαση. Βεβαίως θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε πάρα πολύ στενά αυτή τη δεύτερη φάση. Έχετε δίκιο, έχουν γίνει προσπάθειες, αλλά είναι τόσο μακριά ε, οι στόχοι που έχουμε συμφωνήσει, που θα πρέπει να τις εντείνουμε τις προσπάθειές μας. Ιδίω όσον αφορά τις προσπάθειες, που, τους μάλλον που έχουμε θέσει για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και την ψηφιοποίηση. Και εγώ θα έλεγα από σήμερα ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να βρει έναν τρόπο να αποδεικνύει στους πολίτες ότι τα χρήματα αυτά πιάνουν τόπο, γιατί αυτό, συνάδελφοι, ξέρετε πόσο σημαντικό πρόβλημα είναι Ποιο ξέρει, ποιο το ξέρει ότι πιάνουν ε, τόπο τα χρήματα όλα αυτά που έρχονται από την Ευρώπη. Ε, τίθεται ένα ζήτημα ενημέρωσης των πολιτών όταν γίνονται τόσο μεγάλες ε, επενδύσεις ας πούμε στους σιδηροδρόμους ή επενδύσεις ε, προς την πρόθεση των ποδηλατοδρόμων. Είναι πολύ σημαντικό να το γνωρίζουν αυτό οι πολίτες, να το γνωρίζουν ότι για παράδειγμα κάποιο έργο προς αυτή την κατεύθυνση έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε και εμείς ένα ρόλο να παίξουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Για αυτό το τελευταίο. Θα ήθελα να τονίσω ότι και εμεί βρισκόμαστε στην υπηρεσία σα. Δηλαδή, ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να συνεργαζόμαστε χέρι-χέρι. Κάθε φορά που υπάρχει μια νέα προκήρυξη εκδήλωση ενδιαφέροντο, ε, ερχόμαστε και σα την παρουσιάζουμε, αλλά όπω είπαμε, ε, ήδη έχουμε πολλά 55 έργα, τα οποία πολλά από αυτά βρίσκονται στις εκλογικές σας περιφέρειες. Οποτεδήποτε μας το ζητήσετε, εμείς μπορούμε να σας δώσουμε πληροφορίες για αυτά από την πλευρά της Επιτροπής και είμαστε και στη διάθεσή σας για να μπορέσετε εσείς να δημοσιοποιήσετε, να περάσετε στους πολίτες τι συμβαίνει. Ό,τι στοιχεία θέλετε για να είναι ξεκάθαρη αυτή η επικοινωνία. Ε, Βρισκόμαστε λοιπόν στη διάθεσή σας για να ε, υποστηρίξουμε, να βοηθήσουμε σε αυτή την προσπάθεια δημοσιοποίησης και επικοινωνίας. Πρόεδρο, ευχαριστούμε. Κύριε Ούτερ, σας ευχαριστούμε ε, και για αυτή την πολύ σε καλό κλίμα ανταλλαγή απόψεων που θα συνεχιστεί, είμαι σίγουρη. Μπορούμε εμείς να συνεχίσουμε με την ημερήσια μας διάταξη και να περάσουμε στην παρουσίαση της έκθεσης για τον υπερτουρισμό, τον αντίκτυπό του και πιθανές ε, πολιτικές λύσεις ε, για την αντιμετώπιση του φαινομένου. Δεν θα πρέπει να υποτιμούμε ή να παραγνωρίζουμε, να μην, να μην αντιλαμβανόμαστε σωστά ποιος ακριβώς ε, όρο χρησιμοποιούμε. Ο υπερτουρισμός ορίζεται στην έκθεση αυτή ως μια κατάσταση κατά την οποία έχουμε ένα ξεπέρασμα όλης της δυναμικής μιας συγκεκριμένης περιοχής ή σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Θα ήθελα να ζητήσω από τους συναδέλφους που θέλουν να μιλήσουν μεταξύ τους να βγουν από την αίθουσα. Ευχαριστώ. Έλεγα λοιπόν, ο υπερτουρισμός δημιουργεί προβλήματα επειδή ακριβώς ξεπερνέται το όριο της, που μπορεί να αντέξει μια περιοχή, μια περιοχή σε μια χρονική περίοδο από φυσικής άποψης, από οικολογικής άποψης, κοινωνικής, οικονομικής ή ψυχολογικής. Έγινε λοιπόν μια μελέτη προκειμένου να έχουμε προτάσεις για πολιτικά μέτρα που θα μπορούσαν να ληφθούν για την αντιμετώπιση του φαινομένου. Καλωσορίζω τον κύριο Πολ Πέτερς. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας εδώ, που είναι καθηγητής για τον βιώσιμο τουρισμό στο Πανεπιστήμιο της Μπρέντα και επίσης τον κύριο Κλόντιο Μιλάνο, καθηγητή της, ε, στο, στο τομέα της διαχείρισης του βιώσιμου τουρισμού στο Πανεπιστήμιο της Λέιντα και καθηγητή ανθρωπολογίας στο Πανεπιστήμιο της Βαρκελόνης. Θα σας δώσω έξι λεπτά στον καθένα να ζητώ συγγνώμη, ξέρω ότι είναι πολύ πιεστικό αυτό. Αλλά το βασικό ερώτημα που θα πρέπει όλοι να έχουμε στο μυαλό μας είναι πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα του υπερτορισμού. Έχουμε ήδη πόλεις, τις οποίες οι κάτοικοι διαμαρτύρονται και λένε δεν θέλουμε πια να βλέπουμε τουρίστες. Θα πρέπει λοιπόν να μην υποτιμούμε τα προβλήματα τα περιβαλλοντικά που δημιουργούνται εξαιτίας του υπερτουρισμού. Επίσης δεν θα πρέπει να υποτιμούμε και τον οικονομικό αντίκτυπο. Ε, γιατί οι περιοχές οι οποίες έχουν πληγεί από το φαινόμενο του υπερτουρισμού έχουν πολλαπλά προβλήματα να αντιμετωπίσουν. Κύριε Πέτρας, κύριε Μιλάνο, έχετε το λόγο. Κύριος Πέτρας, σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μας δίνετε να σας παρουσιάσουμε την εκθεσία αυτή. Η μελέτη έγινε το καλοκαίρι του 2018. Έχουν υπάρξει λοιπόν κάποιες εξελίξεις που ίσως να μην συμπεριλαμβάνονται στην εκθεσή μας. Το περιεχόμενο της παρουσίας μας, έχει ως εξή. Αρχικά θα ξεκινήσουμε με μια εισαγωγή κάποιο ορισμό, μια γενική ε, εικόνα του προβλήματος του υπερτορισμού στην Ευρώπη, ε, μεθοδολογία της μέτρηση του φαινομένου και τα αποτελέσματα αυτή. Θα δώσουμε επίση και κάποιε μελέτε περιπτώσεων και ιστάντης και στο τέλος κάποια συμπεράσματα και προτάσεις, ε, συστάσεις προς την Επιτροπή Μεταφορών. Εισαγωγικά να σας ενημερώσω ότι ο σκοπός της μελέτης ήταν να συλλέξουμε πληροφορίες να συλλέξουμε πληροφορίε για την πολιτική που ακολουθείται, βέλτιστε πρακτικέ, καθώ επίση και για τον αντίκτυπο του υπερτορισμού, τρόπου με του οποίου μπορεί να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο, ε, είναι πολύ σημαντικός ο ορισμός του φαινομένου, γιατί υπάρχουν πολλές μελέτες που έχουν γίνει, που χρησιμοποιούν διαφορετικούς ορισμούς. Χρειάστηκε λοιπόν να καταλήξουμε εμείς ένα δικό μας που, που να του συνθέτει και είναι αυτός που βλέπετε τώρα στην οθόνη. Ο υπερτουρισμό περιγράφει μια κατάσταση στην οποία ο αντίκτυπος του τουρισμού ξεπερνάει τα φυσικά, οικολογικά, κοινωνικά, οικονομικά, ε, ε, ψυχολογικά και, ή και πολιτικά κατόφλια, οι δυνατότητε μια περιοχή. Βεβαίω αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά γιατί δεν είναι ότι υπάρχει υπερτουρισμός αν ξεπεραστούν όλα αυτά τα όρια αλλά ξεπεραστεί και μόνο ένα. Και υπάρχουν διάφορες ε, ε, υπάρχουν αρκετές διαφορές μεταξύ των διαφόρων μορφών. Αν δούμε τις αιτίες. Τις τελευταίες ε, δεκαετίες έχουμε δύο εξελίξεις που είναι πάρα πολύ σημαντικές. Η πρώτη είναι ότι οι μεταφορές στον τομέα του τουρισμού έχουν γίνει πολύ φτηνές και πολύ γρήγορες. Κυρίως μέσω πτήσεων χαμηλού κόστους ε, σε αερομεταφορές, αλλά και οι διπηρεωτικές ε, διασυνδέσεις έχουν γίνει πάρα πολύ φτηνές. Αυτό σημαίνει ότι κάθε προορισμός, κάθε χωριό στην Ευρώπη είναι μια δυνητική αγορά για ολόκληρο τον κόσμο. Ε, ήταν πολύ τοπικό το φαινόμενο, αλλά έχει επεκταθεί δυνητικά βεβαίως. Η δεύτερη σημαντική εξέλιξη αφορά την τεχνολογία, ψηφιακές ε, πλατφόρμες, ε, κοινωνικά μέσα. Αυτό το οποίο συμβαίνει είναι ότι βασικά κάνουν κάποια μέρη μόδα. Δηλαδή αν κάποιος προορισμός εμφανιστεί λίγο σε ενδιαφέρον, ε, ξαφνικά γίνεται ο πιο ενδιαφέρον ε, προορισμός στην Ευρώπη. Και αυτή η μόδα σε συνδυασμό με άλλους ε, παράγοντες οδηγεί σε κάποιους λίγους προορισμούς να έχουν τεράστια τουριστική κίνηση. Δηλαδή υπερτουρισμό βεβαίως έχουμε την διάδοση των μη ρυθμισμένων καταλήμματων όπως το Airbnb και το πρόβλημα είναι ότι ενώ χρειάζεται περισσότερη διακυβέρνηση τα συστήματα αυτά δεν ε, ε, ρυθμίζονται, δεν πληρώνουν φόρο και δεν υπάρχουν ρυθμίσεις. Οπότε μπορούν να μην υφίστανται καμία ρύθμιση. Γενικά έχω... έχουμε δημιουργήσει ένα μοντέλο, το βλέπετε εδώ πέρα, υπάρχει και στην έκθεση και μας λέει απλά ότι εάν ο αντίκτυπος του τουρισμού ξεπεράσει τις δυνατότητες ε, κατά κάποιον τρόπο, τότε ε, μιλάμε για υπερτουρισμό. Και βεβαίως ή για διάφορες ε, εξελίξει μετά που ξεπερνούν ε, αυτές τις δυνατότητες. Παγκοσμίω, το 2018 το καλοκαίρι ε, βρήκαμε 105 προορισμούς με υπερτουρισμό ε, εκ των οποίων βρήκαμε 70 στην Ευρώπη. Βεβαίως περισσότερο κοιτάξαμε την Ευρώπη. Δεν, μάλλον δεν ισχύει ότι έχει τους περισσότερους προορισμούς η Ευρώπη ο αντίκτυπος ε, του υπερτουρισμού ε, φτάνει και δημιουργεί υπαρξιακά ζητήματα. Σε κάποιες περιπτώσεις οι κάτοικοι φεύγουν. Ε, μειώνονται κατά 70-80% σε 20 χρόνια και αλλάζει τελείως ένας τόπος λόγω του τουρισμού. Ο υπερτουρισμός έχει κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές πτυχές ε, και ένα σημαντικό θέμα είναι ότι γενικά στον τύπο να μιλάμε για τον ευερτουρισμό στις πόλεις αλλά και τα νησιά, παρακτής περιοχές, ε, περιοχές της υπαίθρου μπορούν να έχουν το πρόβλημα αυτό. Μετά στη μέτρηση του υπερτουρισμού υπάρχει πραγματικά ένα πρόβλημα. Το πρώτο πρόβλημα είναι παραδείγματο χάρη ότι η πυκνότητα των τουρισμών ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο ή ανά κάτοικο διαφέρει τάξη μεγέθους από 4 σε 5 σε 6 ανά προορισμό. Και πάλι θα μπορούσε να είναι ε, κάτι ε, διαφορετικό. Εξαρτάται από την κάθε κατάσταση το είδο, αν υπάρχει κάποια ε, ευπαθή φύση, κάτι τέτοιο. Οπότε είναι μια δυσκολία. Παρ' όλα αυτά, αναπτύξαμε ένα checklist και αν απαντήσει κανείς όλες τις ε, ερωτήσεις, τότε υπάρχει ο κίνδυνος υπερτουρισμού. Και τέλος, τα δεδομένα μας βασίστηκαν στα στατιστικά ΝΑΤΣ ε, 2, γιατί τα ΝΑΤΣ 3 είναι στο επίπεδο Δήμου που δεν υπάρχουν ε, οι δείκτες που χρειαζόμαστε. Οπότε βασιστήκαμε σε περιφέρειες ε, και με βάση την αξιολόγηση κινδύνου βρήκαμε διάφορες περιοχές στους οποίες υπάρχει κίνδυνος υπερτουρισμού παρά το ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουν κάποιους προορισμούς με υπερτουρισμό. Βλέπετε τον κατάλογο εδώ. Βεβαίως υπάρχουν περιφέρειες που έχουν ήδη ψηλό κίνδυνο. Για να σας δείξω τις ε, διαφορές ε, μεταξύ των διαφόρων δικτών. Στα αριστερά βλέπετε την πυκνότητα αναδιανυκτερεύσεις ε, και ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο και βλέπετε στα αριστερά την ένταση διανυκτερεύσεων, δηλαδή ανακάτοικο. Βλέπετε δηλαδή ότι κάποιες περιοχές από πράσινες ε, γίνονται πιο κόκκινες. Οπότε εξαρτάται πολύ από το που βρίσκεται κανείς στην Ευρώπη και ποια είναι τα χαρακτηριστικά της περιοχής. Παρ' όλα αυτά, βρήκαμε κάποιους στατιστικά σημαντικούς δείκτες για τον κίνδυνο υπερτουρισμού που αναφέρονται εδώ στα αριστερά. Παραδείγματος χάρη υψηλό ποσοστό του τουρισμού στο ΑΕΠ, η πυκνότητα του τουρισμού, η ένταση του τουρισμού, η ανάπτυξη των αερομεταφορών. Ε, αυτό είναι ένας ιδιαίτερος παράγοντα κινδύνου. Επίσης ε, το ποσοστό του Airbnb ε, στις συνολικές ε, διανυκτερεύσεις και κλίνες. Δεν βλέπουμε εδώ πέρα τις διάφορες περιπτώσεις που είδαμε, τους προορισμούς που είδαμε στην Ευρώπη, η μεγαλύτερη κύκλη ε, είναι οι μελέτες που κάναμε, τις επιλέξαμε ε, για να έχουμε τουλάχιστον ένα σε κάθε χώρα. Και έχουμε μια ωραία κατανομή μεταξύ πόλεων, υπαίθρου κτλ. Και παρακτήων περιοχών και νησιών. Ε, από τις περιπτώσεις που εξετάσαμε βλέπουμε ότι ο αντίκτυπος εξαρτάται από το είδος του προορισμού, εάν μιλάμε για ύπεθρο ή για φύση. Βεβαίως υπάρχουν ζητήματα οικολογικά στις πόλεις, ε, θα είναι πιο κοινωνικά τα ζητήματα με τους κατοίκους. Επίσης είδαμε τα μέτρα τα οποία ε, λαμβάνονται στους προορισμούς υπερτορισμού και σχετίζονται με την κατανομή των επισκεπτών σε χώρο και χρόνο στο να αλλάξει η ακατάλληλη συμπεριφορά των επισκεπτών, στο να αυξηθεί ε, η δυνατότητα των υποδομών. Ε, ε, Βεβαίω εδώ πέρα δεν υπάρχει κάτι για την αύξηση του ίδιου του τουρισμού. Και τέλος, κάτι άλλο το οποίο μάθαμε από αυτές τις περιπτώσεις είναι ότι δεν υπάρχει κάποια παρακολούθηση των μέτρων ε, του υπερτουρισμού, οπότε ε, τουλάχιστον δεν υπήρχε μέχρι πέρσι. Και κάποια βασικά συμπεράσματα. Τα αποτελέσματα, οι επιπτώσεις ε, μπορεί να είναι πολύ σοβαρές και υπαρξιακές. Βεβαίως εξαρτάται, όπως είπαμε, από τον προορισμό το θέμα της ανάπτυξης που είναι πραγματικά πρόβλημα και όπως είπαμε οι φτηνές πτήσεις σε συνδυασμό με τα κοινωνικά μέσα που συνεισφέρουν σε αυτό και τέλος σχεδόν τέλος κάποιες συστάσεις πρέπει να γίνει πιο συστηματική έρευνα να έχουμε πιο λεπτομερή στατιστικά σε επίπεδο 3 και τέλος είμαστε. Η τελευταία σύσταση, οι άλλε είναι αυτεξήγητες, είναι η δημιουργία μιας task force ε, πανευρωπαϊκής ε, για τον υπερτουρισμό, για να οργανωθεί έρευνα χρειαζόμαστε στατιστικά στοιχεία. Και εμπειρίες από διάφορους προορισμούς. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ μια task force σε ευρωπαϊκό επίπεδο, λέτε, αυτό έχουμε κάνει εδώ ήδη στην Επιτροπή μας. Δημιουργήσαμε μια task force για τον τουρισμό και αυτό το ζήτημα του υπερτουρισμού θα είναι ένα από τα μελήματά της. Κύριε Μιλανό, για 6 λεπτά έχετε το λόγο. Μπορείτε και εσείς να τα ξεπεράσετε λιγάκι αν θέλετε, όπως ο κύριος Πίτερς. <clears throat> Um, good morning. More than... Ο κ. Πίτερ ε, υπογράμμισε τα πιο σοβαρά συμπεράσματα της έκθεσης, οπότε ε, ε, είχα την εντύπωση ότι θα έκανε την παρουσίαση και μετά θα απαντούσαμε σε ερωτήσεις. Όπως είπε πάντως, έχει ήδη περάσει ένας χρόνος και σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχουμε διαπιστώσει αύξηση των κοινωνικών εντάσεων σε σχέση με τον τουρισμό, ως αντίδραση στον τουρισμό. Να συνεχίσουμε, να ξεκινήσουμε τη συζήτηση τότε, κύριε Μαρινέσκο. κ. Μαρινέσκου, ευχαριστώ πολύ γιατί την παρουσίαση είναι πολύ χρήσιμη αυτή η μελέτη για μα για τη βιομηχανία τουρισμού, για όλους. Παρουσιάσατε ένα κατάλογο κινδύνων. Μεταξύ αυτών δεν είδα ε, τον κίνδυνο χειροτέρευση τη ποιότητα των υπηρεσιών. Νομίζω ότι όταν έχετε κανείς πολλούς τουρίστες είναι υπάρχει ο κίνδυνος ορατός να πέσει η ποιότητα. Έτσι λειτουργεί το σύστημα. Το ελέγξατε ή όχι. Και αν το ελέγξατε, μπορείτε να μας πείτε ποια είναι τα συμπεράσματά σας. Και ο, Ευχαριστώ πολύ την, της τους ε, κυρίους που μας έκαναν την παρουσίαση. Δεν θα ασχολιάσω τα πάντα βέβαια, δύο λεπτά μόνο μου δίνετε. Να εστιάσω στο δικό μας καθήκον εδώ ως Επιτροπής. Εμείς πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι αυτοί που λαμβάνουν τις αποφάσεις, ανεξαρτητός επίπεδου, εθνικές κυβερνήσεις, Βρυξέλλες, τοπικές αρχές, οποιοδήποτε και αν είναι αυτοί, θα καταλαβαίνουν, θα καταλάβουν ότι χρειαζόμαστε καλύτερο συντονισμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Χρειάζεται να γίνει μια πρόθεση, ένα marketing σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πλήθη σε πολλά σημεία τη Ευρώπης, ενώ με μια ευρωπαϊκή προώθηση του τουρισμού θα μπορούσαμε να προωθήσουμε και άλλα μέρη στα οποία δεν εμφανίζεται αυτό το φαινόμενο του υπερτουρισμού. Το κοινό θα πρέπει να καταλάβει ότι η Ευρώπη διαθέτει πάρα πολύ πολύ όμορφα μέρη και ο τουρισμός μπορεί να κατανεμηθεί σε περισσότερους προορισμούς. Αυτό όμως χρειάζεται συντονισμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Χρειαζόμαστε στο 7 ετές πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο μία γραμμή προπολογισμού για το βιώσιμο τουρισμό. Αυτό θα μας επιτρέψει να εξασφαλίσουμε αυτές τις κοινέ ευρωπαϊκού επίπεδου εκστρατείες προώθησης του ευρωπαϊκού τουρισμού. Η καινούργια πρόεδρος, κ. Φάντερ Λάιεν, δεν έχει αποφασίσει ακόμα αν κάποιος από τους επιτρόπους θα είναι υπεύθυνο για τον τουρισμό. Ο κ. Τίμερμανς έχει αναλάβει να διαχειριστεί την Πράσινη Συμφωνία και σε πολλά σημεία αυτού του Green Deal υπάρχουν ζητήματα συναφή με τον τουρισμό. Κατά την άποψή μου θα χρειαζόμασταν όμως κάποιον επίτροπο που να εκπροσωπεί τον τουρισμό. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις αρνητικές πτυχές, τις αρνητικές συνέπειες του τουρισμού. Και θα μας επέτρεπε να ακούσουμε και τη φωνή των εμπειρογνωμών και τη φωνή των τοπικών αρχών. Για να εξασφαλίσουμε ότι ο τουρισμός δεν καθίσταται εχθρός του λαού, αλλά αντιθέτως τον εκπροσωπεί. Ευχαριστώ πολύ. Ο κ. Δίαθ. θα μιλήσω ισπανικά. Το πρώτο που θέλω να κάνω είναι να ευχαριστήσω τους δύο καθηγητές για την παρουσίασή τους. Όλοι γνωρίζουμε ότι ο τουρισμός στην Ευρώπη αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις. Την ψηφιοποίηση, τα νέα επιχειρηματικά μοντέλα. Το Thomas Cook είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα μη προσαρμογής. Η βιωσιμότητα, η ανταγωνιστικότητα η προσέλκυση νέων τουριστών και σίγουρα η καταπολέμηση του υπερβολικού τουρισμού που οδηγεί σε μείωση της ποιότητας, σε χειροτέρευση της ποιότητας. Θέλω να ευχαριστήσω λοιπόν τους δύο καθηγητές που συμπεριέλαβαν και τις Βαλεαρίδες νήσους. Ήμουν πρόεδρος των Βαλεαρίδων νήσων για κάποια χρόνια και γνωρίζω πολύ καλά το φαινόμενο. Πάντοτε πίστευα και εξακολουθώ να πιστεύω ότι θα πρέπει να δώσουμε έμφαση στην ποιότητα και όχι στην ποσότητα. Και οι Βαλεαρίδες νήσι είναι πρότυπο ακριβώς γιατί έκαναν πολλές μεταρρυθμίσεις σε κρατικές πολιτικές στις υποδομές τους και συνεργάστηκαν οι αρχές πολύ στενά με τον κλάδο. Ένας κλάδος ο οποίος έκανε πολλές επενδύσεις για τη βελτίωση των εγκαταστασεών τους μια μεγάλη σημαντική προσπάθεια ε, διάδοσης και προώθησης, μια σημαντική προσπάθεια ε, κατανομής του τουρισμού σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα μέσα στον χρόνο, ε, προβολής του πολιτιστικού τουρισμού κλπ. Η Βαλερίδες νήσι δεν είναι το μόνο πρότυπο, βέβαια, αλλά αναπτύσσεται και το φαινόμενο της τουρισμοφοβίας σιγά σιγά σε πολλές περιοχές της Ευρώπης. Ο τουρισμός δημιουργεί εκατοντάδες χιλιάδες θέσεων εργασίας. Γι' αυτό το λόγο δεν θα πρέπει να τον βλέπουμε ως εχθρό αλλά ως ευκαιρία. Έτσι θα πρέπει να τον αναλύουμε, όχι ως απειλή. Προφανώς θα πρέπει να λειτουργούμε με βάση κριτήρια επιλογής, ποιότητας κλπ αλλά είναι ευκαιρία ο τουρισμός. Εμείς ως ε, Ciudadanos, το κόμμα μας δηλαδή, ε, είμαστε αποφασιστικοί. Θέλουμε να αποφύγουμε τον τουρισμό, την τουρισμοφοβία, θέλουμε να αποφύγουμε να ενοχοποιήσουμε τον τουρισμό. Δεν θέλουμε την μείωση του τουρισμού μέσω αύξησης φορολογίας θέλουμε να ενισχύσουμε τον τουρισμό, αλλά τον ποιοτικό τουρισμό, όχι τον ποσοτικό τουρισμό. Τέλος έχω την εξή σκέψη. Πολύ συχνά τον τουρισμό τον αντιμετωπίζουμε ως ένα αεροδρόμιο, ένα εστιατόριο, ένα ξενοδοχείο. Όχι. Ο τουρισμός είναι κάτι πολύ περισσότερο. Είναι μια εμπειρία. Είναι η αίσθηση που αποκτούν οι τουρίστες και επιστρέφουν με αυτή στην πατρίδα τους είναι ένα άθροισμα. Όλο το άθροισμα αυτό είναι μια εμπειρία. Και έχουμε μια ευθύνη όλοι εμείς. Αυτή η εμπειρία θα πρέπει να είναι η καλύτερη δυνατή για τους τουρίστες. Και όπως λέτε και εσείς, θα πρέπει να βασιστούμε στην ποιότητα και όχι στην ποσότητα. Αυτό και τελειώνω ξανά ευχαριστώντας σας και ενθαρρύνοντας μας να εξακολουθήσουμε να δουλεύουμε για αυτό το θέμα. Merci beaucoup, Monsieur Baudiat, Monsieur Koff. Δεν ξέρω πώς διαβάζετε αυτό. Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ επίσης και ο κύριο που μα έδωσε μια πλήρη εικόνα των διαφόρων προβλημάτων που δημιουργεί ο υπερτουρισμό. Πρέπει να σκεφτούμε και τις δύο πλευρές, δηλαδή το ταξίδι προς τον προορισμό και τον αντίκτυπο που αυτό έχει και μετά τον αντίκτυπο στον ίδιο τον προορισμό από τους τουρίστες. Εάν γίνει μια σωστή διαχείριση, ο τουρισμός έχει σημαντικά ωφέλη. Βελτίωση των υποδομών, στον προορισμό, στους τουριστικούς προορισμούς. Δεν είναι δηλαδή όλα αρνητικά όταν προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε την πρόκληση από την εισρωή τουριστών. Αναφερθήκατε στο πρόβλημα που δημιουργεί το Airbnb. Το τονίζω και εγώ, είναι πολύ σημαντικό το πρόβλημα που έχει δημιουργήσει στην αγορά ε, στέγασης σε κάποιες περιοχές, σε μεταξύ των οποίων και το Δουβλίνο, στην Ιρλανδία από που προέρχομαι. Είναι πολύ δύσκολο το πρόβλημα και θα έπρεπε να ληφθούν ε, πρωτοβουλίε σε διεθνέ επίπεδο για την αντιμετώπιση του. Και είπατε επίση ότι και τα κοινωνικά μέσα δικτύωση έχουν αλλάξει. Ότι κάποιοι προορισμοί γίνονται πολύ δημοφιλείς, κάποιοι άλλοι όχι και δημιουργείται μεγάλη πίεση σε ορισμένους από αυτούς. Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω λοιπόν για την συνεισφορά σας στη συζήτησή μας και θα περιμένω την γραπτή έκδοση της έκθεσης αυτής. Πιο συγκεκριμένα τώρα σε ερωτήσεις. Εξετάσετε το ζήτημα της πιστοποίησης, την πιστοποίηση του βιώσιμου τουρισμού. Και πιστεύετε ότι είναι κάτι το οποίο θα μπορούσε να προωθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, να προωθήσει για παράδειγμα ένα κοινό πρότυπο για τον λεγόμενο πράσινο βιώσιμο τουρισμό, που βεβαίω εντάσσεται σε μια γενικότερη αλυσίδα, αλλά ίσως στην έρευνά σας βρήκατε κάποια παραδείγματα που θα ήταν χρήσιμο να δούμε, για να δούμε τρόπους με τους οποίους μπορεί να γίνει η διαχείριση του τουρισμού με μεγαλύτερη ε, φροντίδα στη βιωσιμότητα του. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Κόφ. Κυρία Βιολό. Καλημέρα κυρία Πρόεδρε, καλημέρα και στους συναδέλφους και ευχαριστώ μου δώσετε τον λόγο. Η έρευνα αυτή είναι και ενδιαφέρουσα και ανησυχητική. Μέχρι σήμερα δεν υπάρχει κάποια ευρωπαϊκή βάση δεδομένων για την καταγραφή των τουριστικών ροών εσωτερικών και εξωτερικών. Δεν υπάρχει μια συντονισμένη τουριστική πολιτική. Βλέπουμε λοιπόν απλά το ότι συμβαίνει και βεβαίως ε, δεν μπορούμε παρά να ενθαρρύνουμε την άντληση δεδομένων από το Booking και το Airbnb αφού λείπουν ευρωπαϊκές και εθνικές πολιτικές. Εμείς όμως θα μπορούσαμε να ζητήσουμε μεγαλύτερη διαθεσιμότητα κονδυλίων για άντληση δεδομένων και από τους μεγάλους tour operator. Επίσης ε, προστάθηκε μια task force για τον τουρισμό. Καλώς, αλλά η δική μας Επιτροπή τι κάνει. Η Ευρώπη αυτή τη στιγμή δεν έχει κάποιον ε, αρμόδιο επίτροπο. Η η κυρία Φαντερ Λάιεν δεν έχει πει κάτι σχετικό. Επίσης βλέπουμε διάφορα μέρη στην Ευρώπη, Νάπολη, Κάπρι, Βενετία, Μπρίζ κτλ που βασίζονται στον ε, τουρισμό χωρίς να σκεφτόμαστε τις πιθανές ζημιές στην ε, κληρονομιά, την πολιτιστική και την ε, καλλιτεχνική. Τα δεδομένα επίσης αυτά αναφέρονται στο 2018. Δεν ξέρω λοιπόν αν υπάρχουν νεότερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Η κυρία Κουντουρά έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω τους δύο καθηγητές. Ε, έχουν κάνει μια πολύ καλή προσπάθεια να δώσουν τα προβλήματα τα οποία δημιουργεί ο υπερτουρισμός και σε προορισμούς αλλά και γενικότερα στην αντιμετώπιση του. Ε, ο χειρισμός όμως του φαινομένου χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή γιατί μπορεί να έχει πολύ αρνητική χρειά και να πλήξει σημαντικά ορισμένους προορισμούς και για παράδειγμα το εξώφυλλο της μελέτης σας είναι μια φωτογραφία από τη Σαντορίνη. Πράγμα το οποίο θεωρώ λάθο, διότι ω Υπουργό Τουρισμού τη Ελλάδα τα 4,5 τελευταία χρόνια μπορώ να σα διαβεβαιώσω ότι η Σαντορίνη δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα υπερτουρισμού. Η Σαντορίνη έχει 365 μέρε το χρόνο τουρισμό και οι όποιες φήμες είδαν το φως της δημοσιότητας ήταν δυστυχώς από κάποιους ανεπαρκείς χειρισμούς των τότε ορισμένων τοπικών ε, φορέων έτσι ώστε ε, έπληξαν την εικόνα του νησιού. Είμαι σίγουρη ότι ο στιγματισμός ορισμένων προορισμών χωρίς στοιχεία δεν βοηθάει στην αντιμετώπιση του φαινομένου. Και η αλήθεια είναι ότι έκπληξή μου επίσης προκαλεί η συμπερίληψη της Πελοποννήσου στη ρίστα στη λίστα με τις 15 περιφέρειες που παρουσιάζουν υψηλό βαθμό κινδύνου να παρουσιάσουν φαινόμενα υπερτουρισμού, δεδομένου μάλιστα ότι τα 4,5 χρόνια στην Ελλάδα προσπαθούμε να προωθήσουμε τουριστικά την Πελοπόννησο, γιατί έχει πολύ μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης. Εδώ λοιπόν θέλω να κρατήσω τα συμπεράσματά σας ότι δεν υπάρχουν επαρκή στατιστικά στοιχεία για τη μελέτη του υπερτουρισμού και δεδομένου ότι η μελέτη αυτή ολοκληρώθηκε πριν από ένα χρόνο και ο τουρισμός τρέχει με πολύ μεγάλες ταχύτητες. Και έχετε επίσης εντοπίσει 105 προορισμούς που αντιμετωπίζουν, λέτε, το πρόβλημα του υπερτορισμού, χωρίς όμως να υπάρχουν σαφή κριτήρια. Και αυτό είναι, νομίζω, μία έλλειψη της μελέτης. Προτείνω, λοιπόν, <clears throat> ένα πιλωτικό πρόγραμμα με τη βοήθειά σας, ώστε να γίνει ένα πρώτο βήμα για μια εκτενή καταγραφή δεδομένων και ορισμού των πραγματικών ενδείξεων για την ύπαρξη φαινομένων υπερτουρισμού, διότι το Task Force που προτείνεται δεδομένου ότι όπως είπε και η κυρία, Υπουργό, η κυρία Πρόεδρος έχουμε ήδη στην Επιτροπή μας ε, δημιουργήσει ένα task force που μπορεί να ρυθμίσει αυτά τα θέματα. Ε, δράτω της ευκαιρίας να πω ότι η Επιτροπή μας έχει ζητήσει από την κυρία Φοντερ Λάιεν να έχει και στην ε, Κομισιόν, ο Commissioner, το πορτοφόλιο Transport and Tourism, μεταφορές και τουρισμό. Θα είναι πιο εύκολο και για μας να συνεργαστούμε με την ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θεωρώ ότι η πρόταση που έχουμε κάνει για έναν ολοκληρωμένο ευρωπαϊκό μηχανισμό διαχείρισης είναι η... Ouais, είναι η πιο σωστή, διότι εκτός από τον υπορτουρισμό, ο τουρισμός πρέπει να αντιμετωπίσει ευρωπαϊκά όλα τα προβλήματα της κρίσης, τα ακραία φαινόμενα, τα καιρικά, την κλιματική κρίση, τα ζητήματα μετανάστευσης, ασφάλειας, πτωχεύσης τουριστικών κολοσσών. Νομίζω ότι αυτό θα έπρεπε να το δείτε εκτενέστερα. Ευχαριστώ. Merci Madame Kundura. Alors je vais réduire à 1 minute 30 parce qu'il y en a qui prennent le temps de parole des autres. Tant pis. Θα μειώσω το χρόνο των υπόλοιπων στα 1,5 λεπτό διότι κάποιοι τον υπερέβησαν οπότε ε, δεν έχουμε αρκετό χρόνο. Παρακαλώ έχετε το λόγο κύριος Φλέγκο. Θέλω να ευχαριστήσω και εγώ τους ε, δύο καθηγητές. Ε, έρχομαι από την Ίστρια, ε, την πιο ανεπτυγμένη τουριστικά περιοχή της Κροατίας. Γνωρίζω πολύ καλά τους κινδύνους που δημιουργεί ο τουρισμός. Όσο καλά και να διαχειριστούμε τον τουρισμό, θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και να γνωρίζουμε τον κίνδυνο του υπερτουρισμού, να εστιάζουμε στην ποιότητα και όχι στην ποσότητα. αν, αν πάρουμε το λόγο των τουριστών ε, προς τους κατοίκους, ε, ε, θα έλεγε και θα βγάζαμε το συμπεράσμα ότι η Ισλανδία είναι πρώτη, η Κροατία είναι δεύτερη, η Τσικουετέρε τρίτη και το Ντουμπρόβνικ τέταρτο. Ε, αυτές οι δύο τελευταίες είναι οι δύο πρώτες από πλευράς πόλεων. Ε, α, αλλά ας δούμε λίγο τις λύσεις και όχι τα προβλήματα. Έχουμε τρία στοιχεία εδώ. Πρέπει να αναπτύξουμε τις υποδομές μας, ε, αποχετεύσεις, ε, δρόμους και εκεί θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το, τα, τα ταμεία συνοχής. Στο επόμενο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο θα πρέπει ήδη να δούμε πώς θα καλυφθούν αυτές οι, αυτές οι υποδομές. Δεύτερον, το κράτος θα πρέπει να παρεμβαίνει με μέτρα για την μείωση του κόστους στον τοπικό πληθυσμό, διότι αυξάνεται το κόστος ζωής εκεί πέρα στις περιοχές που υπάρχει πολλής τουρισμός. Τρίτον, θα πρέπει να ενθαρρύνουμε την ψηφιοποίηση. Οι ψηφιακές πλατφόρμες μπορούν να μας βοηθήσουν να χειριστούμε καλύτερα τις ε, κινήσεις των τουριστών και τις τάσεις. Να μειώσουμε τις, την πίεση σε συγκεκριμένους, σε συγκεκριμένους προορισμούς. Ευχαριστώ. Ο κύριος Σκοτ, ευχαριστώ πολύ για τις, ε, σαφείς αυτές, για παρουσίαση. Μακάρι όλες οι παρουσιάσεις να ήταν τόσο σαφείς. Γιατί πραγματικά θα είχαμε αντιμετωπίσει ε, τις κλιματικές απειλές ήδη. Χαίρομαι που η Κομισιόν έχει ε, ασχοληθεί με το θέμα αυτό. Θα μπορούσε η Κομισιόν όμως να δει έναν να δει το θέμα της ε, κλιματικής, ε, του, της κλιματικής απειλής μέσω όλων των συνιστοσών του τουρισμού. Δηλαδή να δούμε πώς όλες οι πτυχές του τουρισμού μπορούν να επηρεάσουν την κλιματική αλλαγή. Θα ήθελα να συνεχίσουμε αυτή τη δουλειά, να συνεχιστεί αυτή η δουλειά, γιατί δεν μπορούμε να συνεχίσουμε στην πεπατημένη. Ο, αριθμός των τουριστών είναι πλέον μη βιώσιμος. Και η αύξηση είναι επίσης μη βιώσιμη. Για να βγάλουμε χρήματα θα παραχωρήσουμε τις ακτές μας, θα καταστρέψουμε περιοχές φυσικού κάλους, που εμείς βέβαια θα τις έχουμε γνωρίσει, αλλά οι επόμενες γενιές δεν θα τις γνωρίσουν κλπ. Ο αστικός τουρισμός είναι πολύ σημαντικό επίσης να, να, το, να τύχει σωστής διαχείρισης. Ε, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πραγματικά πάρα πολύ για την πολύ σαφή σας παρουσίαση. Ευχαριστώ. Πρόεδρος. Κυρία Κουντουρά. κυρία Κουτάγιαρ. Ε, δεν ήταν, το είπατε πολύ σωστά το όνομά μου, δεν πειράζει. Έχετε τόσα πολλά ονόματα να πείτε. Ευχαριστώ πολύ για αυτήν την παρουσίαση, την πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη. Ε, να υπογραμμίσω τα εξή δύο πράγματα. Πρώτον, τη σημασία να υπογραμμίσουμε ότι πρέπει να διαθέτουμε επαρκή στατιστικά στοιχεία στο μέλλον. πολύ συχνά τα στοιχεία τα οποία συλλέγονται δεν λαμβάνουν υπόψη τους καινούριους τύπους ε, του τουρισμού, τους, δεν λαμβάνουν υπόψη όλους τους προορισμούς κλπ. Επίσης, θα σας θυμίσω το δημοψήφισμα που έχει προγραμματιστεί στην Βενετία για τον υπερτουρισμό. Βλέπετε ότι οι τοπικές κοινωνίες αντιδρούν. Όμως τα δημοψηφίσματα και οι δικαστικές αποφάσεις δεν είναι οι πιο κατάλληλες λύσεις. Πρέπει να δούμε και, άλλες, και άλλα παραδείγματα. Να σας ρωτήσω λοιπόν το εξής. Υπάρχουν παραδείγματα τα οποία λάβατε υπόψη στη μελέτη, τα οποία θα, μπορούσατε, θα μπορούσαν να μας βοηθήσουν στον, στην καταπολέμηση του φαινομένου του υπερτουρισμού που δεν περιορίζεται στη Βενετία. Για ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ και για την παρουσίαση. Εδώ πέρα έχουμε ένα θέμα το οποίο αφενός είναι δύσκολο να καθοριστεί και δύσκολο να μετρηθεί κιόλας δεν είναι εύκολη υπόθεση. Πριν έρθω στο ερώτημά μου, θα ήθελα να σας παρακαλέσω να επιλέγουμε προσεκτικότερα τις λέξεις μας, γιατί είναι πολύ σημαντικό το θέμα. Στη χώρα μου είδα τίτλους εφημερίδων που ε, λέει ότι πρέπει να προειδοποιούν ε, ε, ότι έρχονται τουρίστες. Ε, νομίζω δεν θέμε τέτοια πράγματα. Είπατε ότι η αριθμή είναι του 2018 και το είπατε δύο φορές. Ε, και αναρωτιέμαι ποια είναι η τόσο μεγάλη διαφορά, τι έχει συμβεί δηλαδή ε, τους τελευταίους δέκα στο θέμα αυτό. Δεύτερη ερώτηση αφορά το checklist, ε, τον κατάλογο των ερωτήσεων που επεξεργαστήκατε. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω να επεκταθείτε, ειδικά στο πρώτο και στο τελευταίο σημείο της λίστας αυτής. Τι γίνεται δηλαδή αν κάποιος απαντήσει ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόταση και τις συστάσεις. Οπωσδήποτε ο τουρισμός είναι παράγοντα τη οικονομίας, μπορεί να αναπτύξει μια πόλη, ένα χωριό, αλλά πρέπει να γίνει με τρόπο βιώσιμο. Να σας δώσω ένα παράδειγμα, ε, το οποίο δεν είδα στη μελέτη σας. Η μικρή πόλη ονόματι Χάλστατ ε, στην Αυστρία. Την αναφέρω γιατί τα στοιχεία είναι εντυπωσιακά. Έχει 754 κατοίκους και ένα εκατομμύριο επισκέπτες το έτος. 2.326 επισκέπτες ανακάτοικο. Αν το συγκρίνετε με το Σάλτσμπουργκ το οποίο αναφέρατε, εκεί πέρα έχουμε 12 επισκέπτες ανακάτοικο και μόνο 4 ανακάτοικο στη Βιέννη. Το Σάλτσμπουργκ έχει 1,7 εκατομμύρια επισκέπτες. Στο Χάλστατ έχουμε 1 εκατομμύριο. Ε, θέλω λοιπόν να ρωτήσω και να σας παρακαλέσω να κάνετε το εξή να διακρίνετε μεταξύ των μεγάλων διαφορών όπως Ντουμπρόβνικ, Βαρκελόνη, Βενετία, που είναι σημαντικό το θέμα, αλλά να μην ξεχνάμε και του μικρού τόπου γιατί δεν έχουν τον προπολογισμό να αντιμετωπίσουν αυτό το θέμα. Και βεβαίω υπάρχουν και άλλοι προορισμοί μικροί στην Ευρώπη με λιγότερου από 5 ή 10.000 κατοίκους να του δοθεί ένα προπολογισμό και να γίνει ένα έργο γιατί το πρόβλημα είναι παντού το ίδιο. Ε, πρέπει να πω, η αριθμή αυτή είναι εντυπωσιακή. Ο τουρισμός, θέλω να τονίσω και πάλι, είναι ε, πολύ σημαντικός παράγοντας οικονομίας, βοηθάει στην ανάπτυξη, αλλά ε, όταν έχουμε τέτοιους αριθμούς είναι καταστροφικό όταν αντιμετωπίζει κανείς τέτοια κατάσταση. Ευχαριστώ. Κύριε Ολιβιέ, έχετε ένα λεπτό. Πολύ γρήγορα. Χαίρομαι ιδιαίτερα που έχουμε αυτή τη συζήτηση. Είναι ένα πρόβλημα που επηρεάζει πολλές χώρες ανάμεσά τους και η Γαλλία. Είναι το πρόβλημα περίπλοκο γιατί έχει πολλέ, πολλούς, πολλές και επίσης υπάρχουν και πολλές επιπτώσεις και στο φυσικό περιβάλλον και σε άλλους τομείς. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την ανάλυση που κάνατε και για τις προτάσεις που κάνατε. Ωστόσο πιστεύω ότι όποιε όποιες λύσεις θα πρέπει να είναι κατά κύριο λόγο εθνικές. Ε, μιλήσατε για τον τοπικό τουρισμό Ε, εγώ δεν θα ήθελα να υπάρξει μια ελιτίστικη προσέγγιση στον τουρισμό και ο λαϊκός τουρισμός είναι πολύ σημαντικός και πρέπει να προωθείται και για μένα αυτό είναι προφανές. Επίσης αναφερθήκατε στα προβλήματα που δημιουργούν οι ηλεκτρονικές πλατφόρμες, όμως δεν μπήκαμε σε βάθος. Τα προβλήματα αυτά είναι βιτά. Πρώτα απ' όλα ε, έχουμε προβλήματα σε σχέση με τη φορολόγηση θα πρέπει να τεθεί το ζήτημα της φοροδιαφυγής μέσω αυτών των πλατφορμών γιατί θεωρώ ότι είναι σημαντικό και οι επιχειρήσεις αυτές να συνεισφέρουν στα έξοδα που, στα προβλήματα μάλλον που δημιουργεί η λειτουργία τους. Και το δεύτερο ζήτημα είναι με ποιον τρόπο μπορούμε να ε, συνεργαστούμε καλύτερα να τις, ε, να, ε, προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος, να κάνουμε αυτές τις πλατφόρμες να συνεργαστούν προς το δημοσίου συμφέρον. Αναφερθήκατε στις αεροπορικές εταιρείε low cost. Και πρώτο μου ερώτημα λοιπόν έχει σχέση με το ρόλο τους. Θα πρέπει, για παράδειγμα, να βάλουμε κάποιο όριο γιατί αυτή τη στιγμή βλέπουμε να ανοίγουν περιφερειακά αεροδρόμια για να εξυπηρετήσουν μια low cost και μετά από πέντε χρόνια να πάβει να είναι δημοφιλή ο προορισμό, να αλλάζει η low cost την πολιτική τη και το αεροδρόμιο να μην μπορεί να λειτουργήσει. Αυτό το ζήτημα λοιπόν δεν το αντιμετωπίσαμε. Το άλλο ζήτημα που δεν αντιμετωπίσαμε είναι το ζήτημα του των ωκεανών, των θαλασσών. Γιατί και εδώ έχουμε δυσμενή αποτελέσματα, πτώσει μάλλον του τουρισμού. Το βλέπουμε στην ε, Μεσόγειο, όπου με τα κρουαζιερόπουλια, τα οποία δεν είναι απλώ ένα πλοίο, είναι ολόκληρε κατασκευέ, είναι ολόκληρε πολυκατοικίε που μετακινούνται. Ε, μέχρι πού θα συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, δηλαδή μέχρι πού θα δεχτούμε να καταστρέφεται μια φυσικού κάλους περιοχή για να υποδέχεται αυτά τα πλοία και πώς θα προστατεύσουμε τους τοπικούς πληθυσμούς. Και το τελευταίο που τον έφερε και ο συνάδελφος Ολιβιέ, κατά την άποψή μου, στο ευρωπαϊκό επίπεδο θα πρέπει να αναλυφθούν πρωτοβουλίε για να τεθεί ένα πλαίσιο για αυτές τις πλατφόρμες και ιδιαίτερα το Airbnb. Ε, δεν θα μπορέσουν να το αντιμετωπίσουν μόνο στους διάφορε πόλεις οι οποίες πραγματικά έχουν πνιγεί από αυτό τη νέα μόδα. Έχουμε πόλεις στις οποίες οι κάτοικοι αναγκάζονται να μετακομίσουν, να πάνε να μεταναστεύσουν εσωτερικά επειδή δεν γνωρίζουν πια τον τόπο τους. Και συνήθως ξέρετε ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι επιλέγουν μια εταιρεία low cost ε, για να περάσουν 4-5 μέρες στη Βαρκελόνη είναι εκείνοι που έχουν τα λιγότερο οικονομική, ε, τη μικρότερη οικονομική επιφάνεια. Επομένω θα πρέπει να... Και, έρχομαι σε αυτό που είπατε κύριε Φρυγκό. θα πρέπει να προσέξουμε πώς μπορούμε να προωθήσουμε τη χρήση άλλων μεταφορικών μέσων, όπως για παράδειγμα το τρένο ή ακόμα και το ποδήλατο, για να προωθήσουμε έναν τουρισμό πιο βιώσιμο και για εκείνους που δεν έχουν τα οικονομικά μέσα. Και έτσι λοιπόν τίθεται το ζήτημα του βιώσιμου τουρισμού κατά την άποψή μου. Και να προωθήσουμε επίσης και το περπάτημα. Δηλαδή οι τουρίστες τους αρέσει, όπως γνωρίζουμε, να ε, ξεκουράζονται σιγά σιγά, να μην βρίσκονται υπό συνεχή πίεση χρονική. Τώρα, ξέρω, σα υποβλήθηκαν πάνω από 5 ερωτήματα. Θα σα δώσω 5 λεπτά μονάχα για να απαντήσετε. Ε, βέβαια, θα έχουμε στο μέλλον και άλλε ευκαιρίε να συναντηθούμε. Κύριε Πέτρε, θα ξεκινήσετε εσεί. Κύριε Μιλάνο, εσεί. Ελάτε. Οπότε, Ας ε, ξεκινήσουμε από κάτι που πρέπει να είναι σαφές όταν μιλάμε για τον υπερτουρισμό. Όταν μιλάμε για τέτοια ζητήματα αυτά δεν, δεν σχετίζονται πάντα με τον τουρισμό. Γι' αυτό είναι δύσκολο να αναπτύξουμε κριτήρια και να μετρηθεί ο υπερτουρισμός γιατί ο υπερτουρισμός ε, σχετίζεται με τη στέγαση, τις ε, δημόσιες μεταφορές, την ανισότητα των φύλων, ε, την ποιότητα της εργασίας. Οπότε είναι δύσκολο και είναι πρόκληση να εργαστούμε με μια τέτοια Task Force ε, που θα αγγίξει και όλους τους άλλες παράγοντες ε, που επηρεάζουν τον υπερτουρισμό και βεβαίως είναι και ένας οικονομικός παράγων ο τουρισμός και ως οικονομικός ε, παράγων. Αυτό το οποίο βλέπουμε στο επίπεδο των πόλεων, αλλά βεβαίως εκεί δεν είδα μόνο τις πόλεις, είδαμε και τις παρακτίες πόλεις, την Ήπεθρο και τα σχετικά Έχουμε πάει από εδώ και αρκετές δεκαετίες στο να μιλάμε για προορισμούς και μιλάμε για μια διεύρυνση της τουριστικής φούσκας. Γι' αυτό μιλάμε για Νάπολη, Κάπρι, Τσίνκουετερε, οι άλλες πόλεις στη Βόρεια, η Νότια Ευρώπη που δεν ήταν τουριστικές και τώρα υπάρχουν ε, νέες ε, δυνατότητες ε, και υπερτουρισμός. Αυτό το οποίο πρέπει να μας απασχολήσει και να αναλύσουμε είναι να πάμε από ένα αποκλειστικό μοντέλο σε ένα μοντέλο πιο συμπεριληπτικό. Γι' αυτό βλέπουμε ακριβώς κοινωνικές αναταραχές ε, στην Ευρώπη. Ε, κάποιοι το λένε τουρισμοφοβία ε, που λένε τα μίμια. αλλά υπάρχουν κοινωνικές αναταραχές για το πώς επηρεάζεται η αγοραστική δύναμη σε τέτοιους προορισμούς. Όπως σας είπα, έχουμε ιδιωτικοποίηση δημοσίων χώρων, η ρήπανση, τα προβλήματα του περιβάλλοντος, ε, πρέπει να τα δούμε. Βεβαίω, ο τουρισμός φέρνει ανάπτυξη, ναι, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να δούμε το τι αποτελέσματα έχει ε, στο περιβάλλον. Και τώρα μπορούμε να αλλάξουμε, πρέπει να βρούμε άλλες εναλλακτικές ε, για να μετακινούμαστε ανά την Ευρώπη και παγκοσμίω και αυτό είναι το πρόβλημα και η πρόκληση του τουρισμού και του υπερτουρισμού. Δεν μπορούμε να χρησιμοποιούμε πλέον ε, τέτοιους πόλους ε, μανιχαϊκούς ε, ντόπιοι εναντίον τουριστών. Είμαστε ψηφιακοί νομάδες, εργαζόμαστε διεθνώς. Πρέπει να το δούμε λοιπόν διαφορετικά το πράγμα. Να δούμε και το θέμα της κινητικότητας και βεβαίως ε, να έχουμε και ένα καλύτερο τόπο να ζήσουμε ε, με περισσότερη ισότητα και περισσότερη κοινωνική δικαιοσύνη στις ε, πόλεις. Βεβαίως αυτά τα συμπτώματα και οι αιτίε είναι διαφορετικά. Υπάρχει και μια παροιμία κινέζικη που λέει, αν μου επιτρέπετε να την παραφράσω, είναι σαν τη φωτιά. Μπορείς είτε να μαγειρέψεις είτε να κάψεις το σπίτι σου. Βεβαίω λοιπόν είναι ένα οικονομικό παραγνωτουρισμό, αλλά πρέπει να δούμε τα ζητήματα αυτά του υπερτουρισμού που επηρεάζουν την ποιότητα ζωής ε, ε, πολλών ευρωπαϊκών ε, πόλεων και προορισμών. Σας ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα σας ευχαριστώ και για τα καλά σας λόγια. Δεν μπορώ να απαντήσω όλες τις ερωτήσεις, αλλά Α, ήθελα να τονίσω πάλι κάποια πράγματα. Ακούσαμε το χαμηλό κόστος ε, ταξιδιού και μεταφορών που είναι ένας σημαντικός ε, παράγοντας και ο κύριος παράγοντας ε, είναι ότι κανείς δεν συζητάει τις μεταφορές ε, στα ζητήματα του τουρισμού. Πέρα του ότι εντάξει, θα πρέπει ίσως να υπάρχουν περισσότερες υποδομές σιδηροδρομικές ή στα αεροδρόμια, αλλά το πώς εντάσσεται στο συνολικό προϊόν και τι σημαίνει αν παραδείγματο χάρη υπάρχουν ε, διπυρωτικές συνδέσεις αεροπορικές ότι αυτό δηλαδή έχει συνέπειες ε, για τους ε, κατοίκους. Λοιπόν, η ένταξη αυτή των μεταφορών γενικά ε, δεν γίνεται καλά και από τη μεριά των μεταφορών δεν κοιτάνε καθόλου το θέμα της αναψυχής. Ένα άλλο σημαντικό θέμα, τελικά ο υπερτουρισμός είναι ένα θέμα διοίκησης ε, και πρέπει να το δούμε στην μικροκλίμακα. Κάθε προορισμός είναι διαφορετικός. Δεν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει μια συνταγή και αν κάνετε αυτό όλα θα είναι καλά. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχουν ε, τα μέσα ε, διακυβέρνηση. Οι εξελίξεις αυτές όπως το Airbnb, το Uber και οι άλλες σχετικές πλατφόρμες της οικονομία του διαμοιρασμού σημαίνει ότι χάνετε την δυνατότητά σας να διακυβερνήσετε. Αν όλε οι κλίνε κάπου είναι Airbnb, δεν υπάρχει τρόπος να προστατευτούν οι ντόπιοι όσον αφορά αυτό το φαινόμενο. Άλλο ένα σημαντικό θέμα λοιπόν. Και τέλος ε, για το θέμα της ισότητας αναφέρθηκαν οι φτωχοί που ζουν σε μέρη πολύ... με πολλή κίνηση ενώ οι ίδιοι δεν ε, ταξιδεύουν ή αν ταξιδεύουν είναι πολύ τοπικό το φαινόμενο με μέσα βιώσιμα. Αυτοί είναι οι τουρίστες του μέλλοντος αν θέλουμε βιώσιμο μέλλον. Αυτό είναι αν θέλετε το, το μήνυμα που μιλάμε για την ισότητα, την εισοδηματική π.χ. αυτοί που πετάνε από την Αυστραλία στην Ευρώπη πληρώνουν πολύ λιγότερους φόρους από αυτούς που παίρνουν ένα τρένο στην Ευρώπη από τη μια πόλη στην άλλη. Αυτό πρέπει να το σκεφτείτε. Κάτι δεν πάει καλά σε όρους Και αυτή είναι μια άλλη πτυχή λοιπόν που σχετίζεται και με τον υπερτουρισμό. Και αφορά ακριβώς τις μεταφορές χαμηλού κόστους. Μπορούμε να τους ε, συγχαρούμε και να τους χειροκροτήσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους δύο καθηγητές μας. Θα πρέπει να μας βοηθήσετε και στην Task Force για τον τουρισμό που συστήσαμε. Οπότε δεν θα σας αφήσουμε να εξαφανιστείτε. Γιατί κάποια στιγμή θα πρέπει να καταλήξουμε και σε νομοθετικές προτάσεις. Ο τουρισμός του μέλλοντος θα πρέπει να σέβεται και το περιβάλλον και τη ζωή των πολιτών και τις οικονομικές επιταγές να μην καταντήσουμε ζούγκλα. Ευχαριστώ πολύ. Θα τα πούμε στις 2.30 ξανά με την κυρία Βιανκόφσκα, την Επίτροπο, για να εστιάσουμε στις δυσκολίες που έχουν δημιουργηθεί με την υπόθεση Thomas Cook. Ευχαριστώ. Καλή σας όρεξη. Η πρόεδρος ευχαριστεί και τους διερμηνείς. Ευχαριστούμε πολύ.